Euh, Συνάδελφοι, παρακαλώ σταματήστε τις ιδιωτικές σας συζητήσεις. Καθίστε για να αρχίσουμε στο σημείο 1. Επειδή αύριο επίκειται απεργία στην ε, Γαλλία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ε, ε, εν πάση περιπτώσει, επειδή θα ενδέχεται να μην μπορεί να έρθει ο εισηγητής μας, ε, ο, μάλλον ε, ο κύριος Μόντι ίσως δεν θα μπορέσει να έρθει, οπότε αναβάλλεται η εξέταση αυτού του σημείου. Ε, τα πρακτικά ε, εγκρίνονται από τη συνεδρία στη 17η Μαΐου. Σημείο 3. Ανακοινώσει ε, του Προέδρου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ 7 και 8 Ιουνίου Ε, μιλούσαν για το στόχο της κοινωνικής ένταξης και τη μείωση της φτώχειας στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, ούτως ώστε να ε, ξεφύγουν από τη φτώχεια 20 εκατομμύρια ε, άτομα. Από, εγκρίθηκαν αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κάτι σχετικό τώρα πάλι στα πλαίσια των ανακοινώσεων. Ε, ε συναντηθήκαμε με τη Βελγική Προεδρία μαζί με μια αντιπροσωπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασχοληθήκαμε με τις τρέχουσες υποθέσεις. Η υπουργό Απασχόλησης ανέλαβε την δέσμευση και συμφώνησε να οργανώσει άτυπο τριμερή διάλογο γιατί θα γίνει πριν από την πρώτη ανάγνωση Μα διορθώνει η Πρόεδρος πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Ζητήσαμε από τη Γραμματεία να είναι σε επαφή με τη Βελική Προεδρία, ούτω ώστε να οργανωθεί απευθεία ο άτυπο τριμερή διάλογο μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ε, ε, προβλέπεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στην πρώτη σύνοδο του Σεπτεμβρίου, είναι η εβδομάδα της 6ης Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, και χρειαζόμαστε συμφωνία με το Συμβούλιο με, αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Την ε, Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το δίκτυο APN θα ε, διοργανωθεί εκδήλωση για το θέμα της ένδυας. Και προσκαλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας. Ε, ε, μην κάνετε γκριμάτσες λοιπόν όταν παίρνετε το λόγο. Αυτά για το σημείο 3. Ολοκλήρωσα τι ανακοινώσει μου. Περνάμε στο σημείο 4. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φίγκυρέιντο για την ε, εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών για την έκθεσή τη σχετικά με το ρόλο του ελάχιστου εισοδήματο για την καταπολέμηση τη φτώχεια και για την πρόθεση μια κοινωνία χωρί αποκλεισμό στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο, κυρία Φίγκυρέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, Συνεργαστήκαμε με μέλη όλων των πολιτικών ομάδων, με βουλευτές και τους ε, βοηθούς τους. Και τελικά ε, καταλήξαμε σε μια ομάδα ε, συμβαστικών τροπολογιών που δεν τη χάνουν αποδοχής όλων ε, σε όλες τις περιπτώσεις και κάποιες πλευρές τους αναθεωρούνται ακόμη. Θέλω να το πω εξ αρχής ότι υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στη μετάφραση και στις τροπολογίες μάλλον στις διάφορες ε, γλώσσες και στις αρχικές τροπολογίες και στις συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό ε, ε, δυσχεραίνει πολύ το έργο μας. Εγώ είδα πολλά λάθη, ακόμη και στις δικές μου τροπολογίες. Οπότε στον κατάλογο ψηφοφοριών θα δείτε ότι προτείνονται διάφορες αλλαγές. Η συνηθέστερη ε, είναι ε, τα, ε, η διόρθωση, η εξή διόρθωση, ο μέσος όρος εισοδήματος αντί για μέσο εισόδημα. Είναι δύο έννοιες εντελώς διαφορετικές γιατί μιλάμε για 60% του μέσου εισοδήματος κάθε χώρας που πρέπει να είναι το ελάχιστο εισόδημα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Οπότε ε, είναι καταλητική σημασία σε αυτό για να κατανοήσετε την ε, ίδια την έννοια του ελαχίστου εισοδήματος. Κατόπιν, ε, Υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα, έννοιες ε, λεπτές, ε, ειδικά για την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, το είδος εργασίας, φεριπίν, το, τη φτώχεια, την ένδια, τα είδη ανισοτήτων που πραγματευόμαστε και ερμηνεύονται αυτές οι έννοιες διαφορετικά ανάλογα με τη γλώσσα και έτσι δυσχεραίνει τη εξέβρεση συνενετικής λύσης. Έχουμε διορθώσει διάφορα σημεία με τους συναδέλφους ε, ε, στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Φυσικά ε, υπάρχουν λάθη και σε άλλες γλώσσες που δεν μπορούσαμε να διορθώσουμε. Αν έχετε αμφιβολίες, ελάτε σε επαφή μαζί μας ε, για να διαλευκάνουμε όλα αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε σε ε, καλές συμβαστικές λύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει κέρια σημασία για να υποστηρίξει κάποιος μια συμβαστική τροπολογία. Δηλαδή είναι ένα απλό μεταφραστικό λάθος ε, και εμποδίζει αυτό την έγκριση μιας συμβαστικής ε, τροπολογίας. Λοιπόν, η πρώτη συμβαστική τροπολογία δεν θα δημιουργήσει δυσκολίες, είναι απλή. Νομίζω θα την υποστηρίξει η πλειοψηφία των συναδέλφων, αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στην τροπολογία Β, αν και νομίζω το ίδιο ισχύει. Ε, ε, το, η τροπολογία Γ το ίδιο, δέλτα το ίδιο, δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Σίγματα αυτόρα F Υπάρχουν ε, κάποια γλωσσικά ζητήματα, κρίνω όμως ότι τα έχουμε ήδη διευθετήσει μέσα από τη συζήτηση. Δείτε το κι εσείς, δεν ξέρω αν εντοπίζετε κάποια άλλη δυσκολία. Το ίδιο για το άρθρο F. Εδώ μιλάμε για την εφαρμογή της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας της συνθήκης. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μιλάμε για το άρθρο 9 ε, της συνθήκης. Και το βάλαμε σε παρένθεση για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Για την συμβαστική G ε, πάλι δεν θα υπάρχουν ε, αμφιβολίες. Για την H το ίδιο θα είναι εύκολα τα πράγματα. Για ε, το ή το, το ελπίζω θα δούμε. Το ίδιο και για τη γιώτα. Για τη Τζέι. Τα περισσότερα προβλήματα είναι, ε, σχετίζονται με την τροπολογία Κάπα και μη. και εδώ ε, υπήρχαν πολλά μεταφραστικά λάθη, προσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε και πιστεύουμε ότι πλέον είναι ευκολότερα τα πράγματα και υπάρχει ευρύτερη συνένεση. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω, αν εντοπίσετε κάποια δυσκολία, ε, σας παρακαλώ έρθετε σε επαφή μαζί μου για την συμβαστική M θα έλεγα ότι προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε πολλές ε, διαφορετικές απόψεις αλλά και να κάνουμε και μια υπέρβαση αυτό το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας. Ε, δηλαδή, να έχουμε μια συγκεκριμένη έκφανση, να προχωρήσουμε σε, να έχουμε απτά αποτελέσματα ε, του μέτρου Μιλάμε συγκεκριμένα για το σχέδιο δράσης ούτως ώστε να υλοποιηθεί μια ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα στα κράτη-μέλη. Και εκφράζουμε εδώ διάφορες ιδέες που σχετίζονται με τις εθνικές πρακτικές, με τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις και την κείμενη νομοθεσία. ούτω ώστε να έχουμε κάποια ενδεικτικά πρότυπα για, τις, ε, ο, για τους όρους πρόσβασης, παραδείγματος υπηρεσίες, ε, για τα, τις πρακτικές ε, σε εθνικό, σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε επίσης ε, μέτρα αναφοράς για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής καταπολέμησης της στόχιας και για να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση των βελτίστων πρακτικών. Πιστεύω ότι θα ενισχυθεί το κύρος του Κοινοβουλίου ε, αν εγκρίνει ταχύτατα αυτή την πρόταση, το ώστε σε συνεργασία με το Συμβούλιο και όπως μόλις μας είπε και η Πρόεδρος, να σημειώσει πρόοδο. Αυτός ο στόχος μείωσης ε, του ποσοστού ε, φτώχειας κατά 20 εκατομμυρία, γιατί σήμερα μιλάμε για παραπάνω από 85 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ε, πλέον Κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 100, μέχρι και 120 εκατομμύρια ε, άνθρωποι που ζουν κάτω ε, από τα όρια της στόχιας. Οπότε αν δεν έχουμε συγκεκριμένα μέτρα ούτως ώστε να επικουρήσουμε τα κράτη-μέλη ε, στην υλοποίηση συγκεκριμένων προτύπων, Ε, θα βρεθούμε στην δινή θέση όπου θα έχουμε υποσχεθεί διάφορα πράγματα και τελικά δεν θα έχουμε κάνει τίποτα στην πράξη για να ε, ε, επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο. Κατόπιν τροπολογία 1 σας είπα ότι κάναμε την ε, ε, διόρθωση σχετικά με το μέσο όρο εισοδήματος ε, που είναι λάθος και πρέπει να λέμε μέσο εισόδημα. Κατόπιν στην επόμενη συμβαστική τροπολογία δεν θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε μια, ένα προσωρινό κατάλογο ψηφοφοριών και το τονίζω ότι είναι προσωρινός ο κατάλογος διότι ε, εξετάζουμε κάποιες ενδεχόμενες αλλαγές ε, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που κάνουμε εδώ σήμερα και λαμβάνοντας και υπόψη ε, τις απόψεις των συναδέλφων, το ότι πρεσβεύουν οι πολιτικές ομάδες, τόσο ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινώ αποδεκτή λύση. Ευχαριστούμε η κυρία uh, Thank you very much Λίνε. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και για τα όσα κάνατε για αυτό το θέμα. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των τροπολογιών και προσπαθήσατε να επιτύχετε συμβιβασμός. Εγώ ε, πίστευα ότι η αρχική σας έκθεση ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ ισορροπημένη. Εγώ είμαι υπέρ ενός του μισθού σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά θα πρέπει εδώ να σας πω ότι από πλευράς φιλελευθέρων δεν νομίζω ότι ε, η σωστή λύση είναι μια οδηγία πλαίσιο. Γι' αυτό το συμβιβασμό M δεν μπορώ να καταλάβω, διότι στο συμβιβασμό M λέτε για το μηχανισμό που δημιουργείται, κάπου στο μέσο της συμβιβαστικής τροπολογίας λέτε ότι λέει αυτή, ότι αυτή η πρωτολογία θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα πρόγραμμα δράσης για την οδηγία πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα στα κράτη-μέλη. Η ανησυχία μου είναι ότι εάν οι τροπολογίες που ζητούν οδηγία πλαίσιο δεν περάσουν, η συμβαστική τροπολογία με την οποία κατά τα λοιπά συμφωνώ θα είναι πολύ δύσκολο να την υποστηρίξω διότι έχετε μια σειρά από τροπολογίε που ζητούν μια οδηγία πλαίσιο, μετά δεν θα περάσει το θέμα τη οδηγία πλαίσιο και καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην εφαρμογή από εκεί και πέρα. Ρίξτε του μια ματιά και πέστε μου κατά πόσο έχετε και εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση που δεν ε, περάσουν οι τροπολογίε για, το, ε, για την οδηγία πλαίσιο. Πολλά από τα αναφέρθηκαν στους δείκτες για την ένδυα. Αναφερθήκατε σε ένα 6% ε, κατά μέσο όρο εισοδήματος. Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία, νομίζω, στην τελευταία διάσκεψη του Συμβουλίου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές, διαφορετικοί δείκτες. Και από εκεί και πέρα ε, θα μας λένε τα κράτη-μέλη αν χρησιμοποιούν το χ της 100 του μέσου εισοδήματο, αν μιλούν για, το, για τα νοικοκυριά που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη δεν έχουν ψυγεία, τηλέφωνα, ε, τηλεοράσεις ή άλλα αγαθά θα προτείνω στην ομάδα μου να κατοψηφίσει σε αυτό το 16% όχι γιατί είμαι αντίθετη, αλλά γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι διαφορετικοί δείκτες θα πρέπει να εξεταστούν υπό το φως και τη συμφωνία που επετέχθη στο Συμβούλιο και το γεγονός ότι το Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν ε, εισαγάγεται αυτό το 60%, Ε, δεν είμαι βέβαιη ότι όλα τα κράτη-μέλη θα το πετύχουν. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι δυνατόν να επιτύχουμε αυτό το ποσοστό. Ε, κατά τα άλλα δεν έχω πρόβλημα με τις περισσότερες τροπολογίες και τους άλλους συμβασμούς. Ε, μάλλον μόνο με τη τροπολογία M θα έχουμε πρόβλημα ως ε, πολιτική ομάδα και μας ενδιαφέρει κυρίως αυτό το θέμα της οδηγίας πλαίσιο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο η κυρία Φιγκυρέιντο, εκπονώντας ε, την ε, έκθεσή της και κατά την ε, απόπειρα εξέβρεσης συμβαστικών λύσεων Βέβαια, όπως είπε και η ίδια, υπήρξε στενή συνεργασία με πολλούς εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. και η δική μας πολιτική ομάδα συμμετείχε σε αυτή την αναζήτηση ε, ισορροπημένων συμβαστικών λύσεων, τις οποίες φυσικά και θα στηρίξουμε. Όπως ε, θα έχετε καταλάβει, η συμβαστική τροπολογία κλειδί είναι η M. Αυτή σχολίασε εξάλλου τώρα και η κυρία Λίν. Εδώ θα μπορούσαν να... Αυτό το θέμα μάλλον θα μπορούσε να είναι αμφιλεγόμενο, να όταν ε, ομιλούμε για οδηγία πλαίσιο Όπως βλέπουμε σε αυτήν την τροπολογία θα πρέπει να σεβαστούμε τις εθνικές ε, πρακτικές για να έχουμε και ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει την ε, πρόοδο στον τομέα αυτό. Ε, μιλούμε επίση για την ενίσχυση της καταπολέμησης τη φτώχεια στα πλαίσια της πολιτικής 2020. Διαπιστώνουμε την ε, σχετική αποτυχία στον τομέα αυτό της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ε, διαπιστώνουμε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των 92 και η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 δεν επέτρεψαν την εμφάνιση μιας ομοιόμορφης προσέγγισης σε όλα τα κράτη-μέλη ε, σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα, ενώ είναι προφανές ότι μια τέτοια έννοια, το ελάχιστο εισόδημα, μπορεί να ε, αποτελέσει ε, πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Στο ευρωπαϊκό έτος, λοιπόν, καταπολέμησης της φτώχειας έχουμε την αυτή τη χρυσή ευκαιρία για να αναλυφθεί μια σχετική πρωτοβουλία. Τονίζουμε πόσο σημαντικό, πόσο αναγκαίο είναι να υπερψηφίσουν οι συνάδελφοι την συμβαστική μη, διότι μιλάμε για κοινά πρότυπα σχετικά με την πρόσβαση στο ελάχιστο εισόδημα, δείκτες για την αξιολόγηση του ε, ελάχιστου εισοδήματος, δείκτες ε, για την αξιολόγηση των συμπερασμάτων και παρακολούθηση ε, των αποτελεσμάτων συγγνώμη, και παρακολούθηση των βελτίστων πρακτικών. τονίζουμε τη βαρύτητα αυτής της συμβαστικής ε, τροπολογίας και θα υποστηρίξουμε και όλες τις ε, υπόλοιπες συμβαστικές τροπολογίες που συνέταξε η συγγήτρια. Πρόεδρος. Βγήκα για να υποδεχθώ τον καθηγητή Μόντι, ε, αλλά βλέπω ότι έχουν γραφεί πάρα πολλοί ομιλητές στον κατάλογο στο μεταξύ. Κοιτάζω γύρω-γύρω. Μην ανησυχείτε. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά πρέπει να μπει μια τάξη. Θα πρέπει να διακόψουμε τη συζήτησή μας, να ακούσουμε τον καθηγητή ε, Μόντι και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την ησυχία μας για να μην έχουμε χρονική πίεση και να τοποθετηθούν όλοι ε, για ε, τις συμβαστικές τροπολογίες της συγκεκριάς μας. Συμφωνείτε όλοι? Πάρα πολύ ωραία. Καλωσορίσατε λοιπόν ανάμεσά μας, κύριε Μόντι. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών ε, Υποθέσεων ε, ε, σας ε, καλωσορίζει. Εμείς ε, στον τίτλο της Επιτροπής μας δεν έχουμε και τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως η αρμόδια γενική διεύθυνση, αλλά ίσως προκύψει στο μέλλον. Έχουμε πολλές κοινωνικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς, όπως πολύ σωστά είχατε πει στο παρελθόν. θα ε, εκπονηθούν νέες νομοθετικές και μη προτάσεις από πλευράς της νέας Επιτροπής θα είναι σε εγρήγορση φυσικά ε, η Επιτροπή, ούτως ώστε ε, να επιτευχθεί μια ισορροπία και η κοινωνική διάσταση να μην παραγωνιστεί, να μην παραγνωριστεί η σημασία της κατά την οικοδόμηση της ενίας αγοράς. Χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερα ε, που θα κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, ούτως ώστε στην απαρχή ήδη της διαδικασίας να ε, διαπιστώσουμε αν τα δικά σας συμπεράσματα ε, συνάδουν με τα δικά μας ή σε ποιο βαθμό μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη δική σας ανάλυση. Γνωρίζετε την ε, διαδικασία. Σας δίνω ευθύς αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τιμά, που βρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής σας. Είναι πολύ σημαντικό ε, το έργο σας ε, και όταν ήμουν ε, επίτροπος αρμόδιος για τον ανταγωνισμό εσείς ήσασταν πρόεδρος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και χαίρομαι πολύ που ξανασυνεργαζόμαστε και σήμερα. Σα παραπέμπω σε μια συνέντευξη που είχα δώσει στην εφημερίδα Le Monde πριν από ένα χρόνο. Ο τίτλος ήταν απλώς ε, συμφιλίωση της αγοράς ε, και της ε, κοινωνίας για να τονώσουμε την οικονομία. Ο πρόεδρος Μπαρόσο είχε διαβάσει αυτό το άρθρο, αυτή τη συνέντευξή μου και νομίζω ότι και αυτό έπαιξε ρόλο όταν ε, πήρε την απόφαση να μου ζητήσει να εκπονήσω μία μελέτη ε, για την ε, νέα φάση οικοδόμησης της νέας αγοράς. Τα νέα στοιχεία δεν είναι καλοπιστικά. Νομίζω ότι είναι ένα αναπόσπαστο ε, κομμάτι ε, της ε, όλης διαδικασίας ανασυγκρότησης της αγοράς. Αν δεν σας πειράζει να συνεχίσω στα αγγλικά, λέει ο κύριος Μόντι. Νομίζω ότι το θέμα της νέας παρουσίασης της ενιαίας αγοράς σήμερα είναι πολύ πιο προφανό σημαντικό από ό,τι ήταν ε, τον περασμένο Οκτώβριο όταν ο πρόεδρος Μπαρόβοζο αποφάσισε να ξεκινήσει αυτή τη πρωτοβουλία μέσω έκθεσης για δύο επιπλέον λόγους οι οποίοι κατέστησαν σαφείς έκτοτε. Πρώτον, η κρίση του ευρώ και δεύτερον, η φορολογική κρίση που βιώνουν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Η κρίση του ευρώ φυσικά είναι μια κρίση η οποία οφείλεται σε υπερβολικά ελλείμματα και χρέη. Αλλά η κατά την άποψή μου, σε μεγάλο βαθμό η έλλειψη οικονομικής ένωσης. Έχουμε νομισματική ένωση, αλλά εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε να έχουμε οικονομική και νομισματική ένωση. Και επιτρέψτε μου να υπερβάλλω λίγο, λίγο όμως, ότι στην πράξη η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είχε ένα ίδιο ζευκτικό και από εκεί και πέρα επέλεγαν τα κράτη-μέλη. Είχαμε Οικονομική ή Νομισματική Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια Ευρωζώνη που θεωρεί ότι είναι πιο προηγμένη σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διότι έκανε την επιλογή του ενιαίου νομίσματος, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακολουθεί κατά πόδας ε, τα κράτη-μέλη που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ σε θέματα οικονομικής ένωσης, σε θέματα εναγκαλισμού της ενίας αγοράς, επί παραδείγματι. Και κάποια από τα προβλήματα της Ελλάδος, ε, τα υφέρποντα προβλήματα των δημοσίων οικονομικών, έχουν σχέση με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι ενθαρρυντικό για την Ευρωζώνη το γεγονός ότι παρατηρούμε ότι η Ευρώπη εκτός του ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, τα νέα κράτη-μέλη, έχουν περισσότερη οικονομική ένωση, μεγαλύτερο σεβασμό για την ενιαία αγορά, από ότι τα κράτη της Ευρωζώνης. Και γνωρίζουμε εκ πείρας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, ότι το ενιαίο νόμισμα θα είναι σταθερό και θα έχει οικονομική απόδοση μακροπρόθεσμα μόνον εάν συνοδεύεται και από μια καλά υλοκληρωμένη ενιαία αγορά ε, με κινητικότητα μεταξύ άλλων. Επομένως η κρίση του ευρώ κατά με, είναι σημαντική και ε, αυτό αναφέρεται στο τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσής μου για ε, την ε, επανέναρξη της αγοράς. Τώρα η εννέα αγορά ε, το συζητάμε αυτό, κάποια κράτη-μέλη εδώ και κάποια χρόνια έχουν θέματα σταθερο, φορολογικής σταθεροποίησης, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προκύπτει και από κίνητρα για ανάπτυξη που θα προέρχονται από τον προπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Από πού μπορεί να έχει τις πηγές της η ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Από την αποδυνάμωση του ευρώ, αλλά σε μεγάλο βαθμό, σε επίπεδο των 27, κάποιες από τις ελάχιστες πηγές ανάπτυξης θα είναι μεγάλες περαιτέρω βελτιώσεις στην διάρθρωση του ευρώ μέσω πολύ περισσότερης ολοκλήρωσης δηλαδή μέσω περισσότερης ενέας αγοράς. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους θεωρώ ότι η ενέα αγορά είναι περισσότερο απαράτητη από ποτέ στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, εάν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η εννέα αγορά που είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ είναι και η λιγότερο δημοφιλής από ποτέ στις χώρες μας. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Είναι σχιζοφρενική η κατάσταση. Η απάντησή μου στην έκθεση προς τον πρόεδρο Μπαρόζο για την οποία θα έπρεπε να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί όπως θα γνωρίζετε πολλοί από εσά ε, ε, έκανα διαβουλεύσεις με κάθε μία από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και με πολλές από τις επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου. Επομένως, ναι μεν είναι η έκθεσή μου, αλλά μεγάλο τμήμα της έκθεσης ε, είναι ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και με χαροποιεί το γεγονός ότι είμαι εδώ ενώπιόν σας σήμερα. Η θέση που εκφράζεται στην έκθεση είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα αίτια της έλλειψης δημοτικότητας της ενιαίας αγοράς. Είχα ε, διαπιστώσει πολύ πριν από την κρίση ότι υπάρχει μια κούραση σε θέματα ολοκλήρωσης. Ε, βέβαια ε, υπήρχε και όλο αυτό το δράμα για τις υπηρεσίες και την οδηγία για τις υπηρεσίες στο ε, γαλλικό δημοψήφισμα και έτσι προβλήθηκαν κατά κάποιο τρόπο οι διάφορες ανησυχίες και η γενικότερη δυσαρέσκεια που υπήρχε για το θέμα και πέραν της κούρασης αυτής ως προς την ολοκλήρωση ήρθε και μια κούραση της αγοράς. Ε, χάθηκε ε, το πρεστίζ της αγοράς, ε, τουλάχιστον από αγγλοσαξονικής πλευράς και αν δείτε στα επόμενα χρόνια, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα πολιτικό τοπίο Αύξηση της επιτυχίας μικρών ε, ακροδεξιών και ακροαριστερών κομμάτων που το μόνο κοινό που έχουν είναι η απόρριψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και ακόμα και τα μεγάλα κόμματα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς που ήταν η πολιτική μοχλή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, τις τελευταίες δεκαετίες φαίνονται σαν να ε, χάνουν λίγο τον ενθουσιασμό τους για το ευρώ γιατί ακριβώς εμφανίζονται αυτοί οι πολύ ισχυροί ανταγωνιστές. Το μέλλον λοιπόν της ενιαίας αγοράς είναι από γκρίζο έως πολύ σκοτεινό και όχι ρόδινο σε καμία περίπτωση. Επομένως προτείνω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας, να δούμε τι ανησυχίες υπάρχουν, γιατί ανησυχούμε, σε ποιο βαθμό είναι δικαιολογημένες αυτές οι ανησυχίες, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις παιδαγωγικές εξηγήσεις, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει, αλλά να είμαστε και λίγο ταπεινοί και να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ανησυχίες και να δημιουργήσουμε κίνητρα ε, στις ευρωπαϊκές πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Οι κοινωνικές ανησυχίες, διότι εδώ είμαστε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου, και οι ανησυχίες λοιπόν ως προς την απασχόληση και ως προς τα κοινωνικά θέματα, ναι μεν δεν είναι οι μόνες, αλλά είναι μεταξύ των πιο σημαντικών και θα πρέπει ε, να τις ε, εξετάσουμε. Ξέχασα δεν να πω ότι το γεγονός ότι τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζεται το, το γεγονός ότι η Ευρώπη θέλει να είναι μια ανταγωνιστική οικονομία κοινωνικής αγοράς μας υποχρεώνει και πνευματικός να κατανοήσουμε πώς και κατά πόσον είναι δυνατόν να είμαστε η ψηλά ανταγωνιστική κοινωνική αγορά σε επίπεδο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο και ίσως και η πείρα της Γερμανίας με τις οικονομίες κοινωνικής αγοράς από τους καιρούς του Λούντβιγκ Κέραντ είναι το πιο από το παράδειγμα. Αλλά μπορούμε να ξε... πούμε πράγματι ότι ξέρουμε να συνδυάσουμε την ολοκλήρωση αγοράς και την κοινωνική προσοχή σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σαφείς λύσεις και η έκθεσή μου απλώς κάνει μία απόπειρα να υποδείξει κάποιες οδούς για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πολύ συναρπαστικό κατά την άποψή μου μοντέλο. Στην έκθεση θα βρείτε κατά βάση τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι η δημιουργία μιας ισχυρότερης ε, ενίας αγοράς, να τη δημιουργήσουμε εκεί που δεν υπάρχει, για παράδειγμα στις υπηρεσίες ή στα ψηφιακά συστήματα και ούτω καθεξής. Αλλά επίσης πώς να υπάρχει συνένεση για μια ισχυρή ενία αγορά, διότι αλλιώς δεν θα έχουμε ισχυρή ενία αγορά. Και τρίτον, πώς να έχουμε αποτελέσματα και να έχουμε συγκεκριμένα μία έννοια αγορά. Τα τελευταία λεπτά λοιπόν θα τα αφιερώσω σε κάποιες αναφορές ε, στη συνένεση για μία ισχυρότερη νέα αγορά που είναι και οι πτυχές κοινωνικής φύσεως. Σημείο στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα προκειμένου όχι μόνο να επιτύχουμε κάποιους κοινωνικούς στόχους, αλλά πρωτίστως για να συμφιλιώσουμε την αγορά. Το ένα θέμα είναι οι οικονομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων μετά από τις ε, υποθέσεις ε, Ναβάλ που νομίζω ότι είναι στην παράγραφο 3 της έκθεσης και εκεί ε, πρέπει να σας πω ότι είχα κοινέ διαβουλεύσεις με τους επικεφαλείς της Έτου και της Business Europe για να προσπαθήσουμε να βρούμε διόδους για πιθανές λύσεις, διότι ερχόμαστε όλοι σε δύσκολη θέση εάν η ελευθερία της ενιαίας αγοράς φαίνεται ότι δεν συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, ή αντιστρόφως. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλό αυτό για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πολλό δε μάλλον για τα δικαιώματα των πολιτών. Και εδώ υπάρχουν δύο βασικές συστάσεις στην έκθεση. Η μία διευκρινίζει την εφαρμογή της οδηγίας για την ε, απόσπαση των εργαζομένων και τις πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, η διοικητική συνεργασία και οι κυρώσεις στα θέματα της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων και διαμεθοριακών, ε, διαμεθοριακής υπηρεσιών. Και δεύτερον, εάν υιοθετηθούν μέτρα για να ε, δούμε τα θέματα της εφαρμογής της οδηγίας για τις αποσπάσεις των εργαζομένων, να υπάρχει μια διάταξη που να διασφαλίσει το δικαίωμα της απεργίας βάσει του μοντέλου του άρθρου 2 του, Συμβουλίου ε, του, Κανονισμού του Συμβουλίου του 1998, ο οποίος διευκρίνιζε ότι σε αυτό τον κανονισμό, ο οποίος στόχο είχε να ενισχύσει τις ε, δυνατότητες ελεύθερης μετακίνησης των αγαθών θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διασφαλίσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κατόπιν υπάρχει ένα θέμα που γνωρίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ την Πρόεδρο αλλά και πολλούς από εσά φαντάζομαι για τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ενιαία αγορά. Εκεί έχουμε κάποιες βασικές συστάσεις. Πρώτον, να ενισχύσουμε περιττέρω την ευελιξία για τις οικονομικές αποζημιώσεις, να αναθεωρήσουμε τους κανόνες ε, προμηθειών ε, για να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες των αποζημιώσεων, να παρουσιάσουμε μία πρόταση κατά πάσα πιθανότητα βάσει του άρθρου 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας για ένα κανονισμό ο οποίος θα διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε κάποιες βασικές ε, τραπεζικές υπηρεσίες και να εξετάσουμε την περίπτωση για να επεκτείνουμε κατά πάσα πιθανότητα επί τη βάση του άρθρου 14 και πάλι τις ε, καθολικές υπηρεσίες και την παροχή ευρυοζωνικής πρόσβασης σε όλους. Επίσης, στο θέμα των δημοσίων προμηθειών υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να διασκεδάζουν κάποιες ανησυχίες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ε, φύσεως και τέλος υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο γνωρίζω ότι προκαλεί πάθη. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό αυτό. Ε, προκαλεί πάθη στην κυρία Μπερές για τα φορολογικά θέματα. Νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με τα κοινωνικά θέματα. Μπορεί βέβαια σε κάποιους από εμά να άρεσε να δούμε τολμηρές προτάσεις για την εναρμόνιση της φορολογίας ε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει ανάγκη και κατά πόσον είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη σήμερα. Αλλά είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι μια πιο ταπεινή προσέγγιση σε συνεργασία σε φορολογικά θέματα και συντονισμό σε φορολογικά θέματα είναι και απαραίτητη αλλά και εφικτή και μάλιστα για πολλούς λόγους. Και εδώ έχουμε και συγκεκριμένο παράδειγμα. Το 96-97 είχαμε ένα φορολογικό πακέτο το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στο Συμβούλιο Εκοφέν, Εκοφήν και εκεί είχαμε ένα ε, μικρό μεν αλλά πολύ σημαντικό πακέτο φορολογικών θεμάτων και έγινε πρόταση να δημιουργηθεί ένα μέσο για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά, δημιουργώντας ε, μία ομάδα ε, φορολογικής πολιτικής, ε, την οποία θα προεδρεύει ο Επίτροπος Αρμόδιος για φορολογικά θέματα και θα υπάρχει και συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας. Ξέρουμε τα φορολογικά θέματα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Και να κάνουμε εδώ και τη διασύνδεση με τα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ότι ο σύνδεσμος είναι πολύ ισχυρός, διότι εάν θέλουμε να προχωρήσει η ολοκλήρωση της αγοράς, και πιστεύω ότι θέλουμε περισσότερη ολοκλήρωση και όχι λιγότερη, αλλά δεν γίνει τίποτα με τις συνοδευτικές φορολογικές πολιτικές, τότε θα έχουμε ναι με το πιο κινητό παράγοντα παραγωγής που είναι το κεφάλαιο, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται πολύ περισσότερο τον φορολογικό ανταγωνισμό σε σχέση με τον λιγότερο κινητό παράγοντα παραγωγής που είναι η εργασία. Θα έχουμε δηλαδή μια Ευρώπη η οποία θα υποκρίνεται ότι προσπαθεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας αλλά στην πράξη καταστρέφει τις θέσεις εργασίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρνητικό ακριβώς όπως νομίζω ότι είναι αρνητικό αν το γεγονός ότι το συνειδητοποιούμε αυτό θα δημιουργήσει κάποια μέρα ένα συνασπισμό κατά της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ήταν περιεκτικότατη, διεξοδικότατη η παρουσίασή σας και γύρατε τα ζητήματα που ενδιαφέρουν ε, περισσότερο την ε, Επιτροπή μας. Ο κύριος ε, Σέρκας έχει πρώτο το λόγο και μετά ο κύριος Κρίστινσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μόντι, τον Επίτροπο Μόντι. Καταρχάς να σας πω ότι η παρέμβασή σας ήταν ούμονον πολύ ενδιαφέρουσα, ούμονον πολύ χρήσιμη, αλλά και πολύ τολμηρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τρεις διαστάσεις της παρέμβασής σας, διότι πιστέψτε με είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούμε συχνά τόσο απτά επιχειρήματα σαν αυτά που μας παρουσιάσετε εσείς ε, σήμερα, ευρωπαϊκού πολιτικού χαρακτήρα, αναφερόμενο στην οικονομία με όρους πολιτικής οικονομίας, ε, οικονομίας πολιτικής συζήτησης, συνένεσης, αναζήτησης διεξόδων για να ενισχύσουμε την Ευρώπη και να μην ε, εξαρτώμεθα μόνο από την ε, διάσταση του εμπορίου. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς είναι προφανές ότι στην έκθεσή σας Έχουμε πολλά χρήσιμα στοιχεία για να δημιουργήσουμε αυτή την ε, διευρωπαϊκή συνένεση. Το πρόβλημα είναι ότι η νέα αγορά σήμερα είναι αντιμέτωποι με μια αγορά πολύ ευρύτερη από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και εδώ έχουμε δύο πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε όχι μόνο συνένεση σε κανόνες ε, και συμβιβασμούς ε, σε επίπεδο 27 κρατών μελών, αλλά κατά πάσα πιθανότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Στην εσωτερική αγορά τη δημιουργήσαμε στη δεκαετία του 80-90 ε, με μια οικονομία που τα χρηματοδοτικά θέματα είχαν πολύ λιγότερη σχέση ε, από ό,τι σήμερα πλέον αυτά τα θέματα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα και επιβάλλονται κάποιες προϋποθέσεις που στα υπόλοιπα θέματα της οικονομικής πολιτικής γίνονται πεδαριώδη θέματα, διότι σε ένα βράδυ μία τράπεζα μπορεί να κάνει μία, ένα συνασπισμό κατά μιας χώρας και να καταστρέψουν πέντε χρόνια ε, προπολογισμού και προκλήσεων στον προπολογισμό. Ε, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το χρέος που θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ε, δεκαπλάσιο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Αυτή η διάσταση λοιπόν, η οποία είναι πέραν της Ευρωπαϊκής Συνένεσης, που απαιτεί ε, μία διάσταση του 2020 και πώς προκύπτει από την εκθεσή σας, τι διέξοδοι υπάρχουν, διότι νομίζω ότι αν δεν βρούμε λύσεις, ε, ε, ουσιαστικά έχουμε το γιοφύρι της άρτας. Εμείς το λιμερί και το βράδυ γκρεμίζεται. Εκτιμώ την παρέμβασή σας. Ε, τα ίδια πράγματα με ανησυχούν και εμένα, αλλά έχουμε μια οικονομία όπου η μάχη για την παραγωγικότητα και, τον, ε, και την ανάπτυξη είναι η βασική πρόκληση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ευρωπαϊκά θέματα όταν δεν υπάρχει και μια συνεκτική διάσταση που θα μπορούμε να... Ε, υπερασπιστούμε και προς τα έξω και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε η Ευρώπη να μην είναι ένα νησί απομονωμένο δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα να έχουμε μια ζούγκλα στην οποία δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει μόνο το κέρδος με κάθε μέσο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστενσεν και ο κύριος Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μόντι για την παρουσίαση της νέας στρατηγικής αυτής για την εσωτερική αγορά. Δεν θα πρέπει βέβαια να ενθουσιαστούμε πολύ νωρί, αλλά μου φαίνεται πολύ θετικό το ότι θέλει να πετύχει ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη κινητικότητα ε, αγαθών ε, και κεφαλαίων και την ελεύθερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Χαίρομαι λοιπόν ε, που αποφασίσατε να συντάξετε το άρθρο αυτό για την Λεμόντ, το οποίο διάβασε ο ε, Επίτροπος Παρόζο και ε, τον οδήγησε στο να δημιουργήσει τη στρατηγική αυτή. Μία από τις θεμελιώδεις λήθους της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι η εσωτερική αγορά και αν θέλουμε οι πολίτες να δεχτούν την εσωτερική αγορά, είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιους σωστούς κοινού κανόνες και ένας από αυτούς θα είναι ότι αν ε, μετακινείται κανείς από μια χώρα σε άλλη για να εργαστεί θα πρέπει να εργάζεται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στη χώρα στην οποία φτάνει κανείς. Και το δικαστήριο ξαφνικά θεώρησε ότι πρέπει να, να οργανώσουμε διαφορετικό τρόπο τα πράγματα αυτά και γι' αυτό ε, ε, είχαμε αυτές τις τέσσερις ε, αποφάσεις για την ενιαία αγορά, Λαβάλ, του Λουξεμβούργο και τις άλλες δύο. Και γι' αυτό χαίρομαι που λέτε ότι εξετάζοντας τους νέους κανόνες στην εσωτερική αγορά και με την οδηγία για τις υπηρεσίες που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου πέρσι, την συνθήκη της Λισαβόνας που επίσης τέθηκε σε ισχύ και την ε, οριζόντια κοινωνική ρήτρα. Αυτά ίσως ήδη έχουν αλλάξει κάπως ε, την ε, νομολογία του δικαστηρίου και θα ήθελα να το εξηγήσετε αυτό περαιτέρω. Πρέπει να φροντίσουμε οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς να μην υπερισχύουν των κανόνων στην ε, αγορά εργασίας ε, και στο δικαίωμα προσφυγής. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα στις βόρειες χώρες, γιατί για παράδειγμα η Σουηδία και η Δανία δεν έχουν βασικό μισθό, ελάχιστο μισθό στους νόμους τους ή στις συλλογικές συμβάσεις ή κοινωνικοί εταίροι εποπτεύουν την αγορά εργασίας στην στις χώρες αυτές ε, και ε, έχουμε λοιπόν μόνο το δικαίωμα προσφυγής ε, για να, λυθού, για να, για να λυθούν ενδεχόμενα προβλήματα. Θα είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει για παράδειγμα από την οδηγία για τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σέρτζιο Κοφεράτη και μετά, κύριε Επίτροπε, να απαντήσετε στις πρώτες ερωτήσεις και θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί καθηγητά, συμφωνώ μαζί σας ότι πέρασε πολύ καιρό από τότε που ξεκινήσατε να εκπονείτε το έγγραφο που σας ζητήθηκε και προέκυψαν τέτοιες αλλαγές που ε, ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερα κάποιες από τις ενδείξεις σας. Κάποιες ε, φτάνουν ε, μέχρι και την πρόληψη, κατά την άποψή μου. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, το γεγονός ότι στην έκθεση μας αναφέρατε και εντάχει τη λογική σας. Λέτε ότι πρέπει κατά απογόντως να περάσουμε στη φορολογική εναρμόνιση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, έχοντας ως στόχο να δημιουργηθεί μια αγορά στην οποία δεν θα υπάρχουν ανισότητες και ανισορροπίες και για να ευνοήσουμε την ανάπτυξη, διότι η βασική συζήτηση στην Ευρώπη για μας σήμερα είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει αυτή η ιδέα της εξυγίανσης και ταυτόχρονα δεν αναφέρονται κάποιες αποτελεσματικές και αξιόπιστες γραμμές ανάπτυξης αυτό όσον αφορά τα θέματα της συνένεσης ε, για την οικονομική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κάθε χώρας θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα δεδομένου ότι σε αυτές τις δράσεις εξυγίανσης ε, αναπόφευκτα υπάρχουν κάποιες προσδοκίες και κάποιες προϋποθέσεις ε, για την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Όταν όμως γίνεται εναρμόνιση, εναρμονίζονται ναι μεν και οι αρετές αλλά και κάποια ε, τροτά σημεία. Όσον αφορά λοιπόν την φορολογική πολιτική, δεν είναι λογικό το γεγονός ότι πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια φορολογική πολιτική που δεν ευνοεί τις επενδύσεις. Δηλαδή οι επενδύσεις θεωρούνται πολύ συνηθισμένες δραστηριότητες και παραδόξως έχουν ε, ε, μεγαλύτερα φορολογικά ωφέλη, ε, που έχουν να κάνουν με την αγορά ή τη μεταβίβαση ε, χρηματοπιστωτικών ε, μέσων, προϊόντων. Μήπως εσείς ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στην ε, φορολογική πολιτική, σε αυτό που θεωρείτε, θεωρούμε ότι αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης και αυτό που θεωρείτε πολύ συνηθισμένη δραστηριότητα. Όσον αφορά τώρα την οικονομική ελευθερία και τα δικαιώματα των ανθρώπων, θα ήθελα να προσθέσω στις πολύ σημαντικέ παρατηρήσεις που κάνατε ε, για την ελευθερία της απεργία και το δικαίωμα του απεργή, θα ήθελα να αναφερθώ και στην ελευθερία οργάνωσης. Δεν έχουμε κάποιες ε, τρομακτικέ υποθέσεις που αφορά την ε, ελευθερία κάποιου να οργανωθεί όταν εργάζεται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέτουν την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σε μια επιχείρηση ως αντίθετη με τη συλλογική εκπροσώπηση. Και είναι προφανές εδώ ότι υπάρχει ένα φιλοσοφικό ρεύμα με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν αλλάζει καθόλου την ουσία στο οποίο θα ήθελε ε, να υπάρχει ε, μία αποκλειστική σχέση μεταξύ επιχείρησης και ατόμου, αποκλείοντας κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα της λογικής εκπροσώπησης. Είναι μία μορφή υποχώρησης, η οποία όμως φαίνεται να επανεμφανίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια μέρημνα και νομίζω ότι η αρχή της μέρημνας εδώ θα πρέπει να υιοθετηθεί ε, για να μην βρεθούμε ενώπιον υποθέσεων που μπορεί να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Uh, I would like first of all to... Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους τρεις βουλευτές που πήραν το λόγο μέχρι στιγμής για την μεγαλόψυχη εκτίμησή τους για τη δουλειά μου. Κύριε Σέρκας, νομίζω ότι η παγκόσμια διάσταση, όπως τονίσατε, είναι ε, αποφασιστικής σημασίας. Εάν θεωρήσουμε την εσωτερική αγορά όπως την ανέπτυξε ο Ζακ Ντελόρ πριν ε, ακριβώς 25 χρόνια με μια λευκή ανάπτυξη, με, με, συγγνώμη, με μια με μια λευκή βίβλο που, ε, που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ίσως η σημαντικότερη διαφορά τα τελευταία 25 χρόνια είναι ακριβώς το παγκόσμιο πλαίσιο που δεσπόζει στην σχετικά μικρή δική μας εσωτερική αγορά. Αναφερθήκατε σε αρκετές πτυχές της παγκόσμιας αυτής διάστασης. Προσπάθησα στην έκθεσή μου να το λάβω αυτό υπόψη. Και πρόκειται για εργοτάξιο όπου θα πρέπει η Ευρώπη να προσπαθήσει να κάνει περισσότερα με τις πολιτικές της. Η... κρίση και όλοι περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τα αποτελέσματα της έκθεσης της ε, σχετικής επιτροπής. Η κρίση αυτή λοιπόν ε, έχει αναπτύξει το ενδιαφέρον του κόσμου, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου για πολυμερείς μορφές διακυβέρνησης ε, που αρχικά ε, είχαν εφευρεθεί εδώ στην Ευρώπη και ο Ζαν είχε εφεύρει την διακυβέρνηση της ε, παγκοσμιοποίησης, τη διακυβέρνηση σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις αξίες και τους κανόνες που έχουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η αποδοχή από την Ασία, από την Αμερική αυτών είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν την κρίση, διότι ακόμα και αυτές οι χώρες δεν πιστεύουν πια ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς πολυμερή διακυβέρνηση. Ε, το G20, το G20 για παράδειγμα είναι ένα γέννημα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε η Ευρώπη να μπορέσει να υποβάλει δυναμικά ε, τους κανόνες αυτούς ε, στο παγκόσμιο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται και από την ε, υγεία της Ευρωπαϊκή Οικονομία, την ανταγωνιστικότητά τη. Μακροπρόθεσμα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε και τα δύο. Από τη μία την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι ίσες και ταυτόχρονα να καταβάλουμε προσπάθειες να, ε, έχουμε, ε, ε, να πετύχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού με παγκόσμια πρότυπα. Και, όπως γράφω στην έκθεση, όσον αφορά τους κανόνες για την κρατική ενίσχυση και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Ξέρω ότι του χρόνου η Γαλλία θα προεδρεύει και στο G8 και στο G20. Η Γαλλία είναι πιθανότατα η χώρα που περισσότερο από οποιονδήποτε επιθυμεί η διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο να βασιστεί στο πρότυπο της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι πολύ σημαντικός. Ε, νομίζω ότι ε, ε, ο δημοσιονομικός έλεγχος θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά πολύ σημαντικό για μια ισορροπημένη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ε, οι σχέσεις ε, κρατικών ενισχύσεων ε, με τις επιχειρήσεις κλπ. Και γιατί να μην εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να προωθήσουμε το την παγκόσμια αυτή ατζέντα. Κύριε Κρίστενσεν, ξέρω ότι αναφέρατε δύο χώρες, τη δική σας και τη Σουηδία. τα η συνέπειες για τους ε, εργαζομένους σε απόσπαση είναι σημαντικές στις χώρες αυτές. Ε, δεν μπορώ να πω πολύ περισσότερα από όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση, αλλά ο Λάσλο Άντορ, ο αρμόδιος επίτροπος, βρίσκει πολύ χρήσιμο στους συλλογισμού αυτούς ε, και αυτό με, το, βρίσκω ενθαρρυντικό. Είχα μια συζήτηση μαζί του σήμερα, ξέρω ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την Επιτροπή σας και ελπίζω ότι οι μέθοδοι αυτοί που εντοπίζονται στην έκθεση ε, θα βοηθήσουν τον Επίτροπο να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική. Κάτι που ελπίζω ότι θα ισχύσει και για άλλα μέρη της έκθεσης, διότι αυτή τη στιγμή η έκθεση βρίσκεται στα χέρια της Επιτροπής από τη μία, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και θα πρέπει ε, να ε, αποκτήσει ζωή. Κύριε Κοφεράτη, νομίζω όπως και εσείς και σας ευχαριστώ για τη καλά σας λόγια. Θεωρώ λοιπόν ότι ο συντονισμός, αν όχι και η εναρμόνιση σε φορολογικό επίπεδο είναι ένα σημαντικό βήμα και το θέμα της ανάπτυξης, η διάσταση της ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί τη βάση αυτού του συντονισμού, ο ρόλος της ανάπτυξης, της απασχόλησης και του περιβάλλοντος, ε, της ε, καταπολέμησης αλλαγής του κλίματος. Και εντός αυτού μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Δεν το εμβάθυνα αρκετά βέβαια στην έκθεση, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα φορολογικά συστήματα όσον αφορά σε επενδύσεις. Εγώ ήμουνα πάντα υπέρ και θεωρούσα ότι εντό εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στι δημόσιε επενδύσει και όχι στι δημόσιε δαπάνε. Στο θέμα τη ελευθερία τη απεργία την οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε ε, και για τι τέσσερι ελευθερίε τη ενίας αγορά. το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση ε, κυρίως για τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Δεν το είχα σκεφτεί, ε, βέβαια εσείς με την πείρα που έχετε και με την ευαισθησία σας η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μου δεν είχα σκεφτεί αυτή την πτυχή ε, όχι μόνο την ελευθερία του απεργήν αλλά και την δημιουργία ε, οργανώσεων εντός ε, του εργασιακού δηλαδή την εκπροσώπηση των εργαζομένων Επαναλαμβάνω, δεν έχω εμβαθύνει σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σας. Εάν η ενιαία αγορά θεωρηθεί ο δούριος ύπος ε, για την επίθεση στην ελεύθερη οργάνωση σε αυτές το επίπεδο σχέσεων, πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η ενιαία αγορά θα αντιμετωπίσει ε, κάποια εχθρικά μέτωπα και σας ευχαριστώ πολύ που μου το επισημάνατε. Ε, ευχαριστώ. Άλλους τρεις ομιλητές έχουμε. Ε, εποφελούμε από την απάντηση που δώσατε στον κύριο Κομφεράτη για να τονίσω και εγώ αυτό το σημείο. Γνωρίζετε ότι Είμαστε επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της δράσης ε, του Ταμείου Αλληλεγγύης. Και τις τελευταίες εβδομάδες μας απασχολεί το θέμα της εταιρείας ε, Dell. Ε, είναι εμβληματική αυτή η εταιρεία. Τέλος πάντων, έχει πολλά σημαντικά στοιχεία αυτή η υπόθεση. Δεν θα μακρηγορήσω. Μιλάμε για ε, μετατόπιση δραστηριοτήτων στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην Ιρλανδία είχε πάρα πολλούς μισθωτές, ε, διότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης αφορούσε πάνω από χίλιους μισθωτούς. Ε, γι' αυτό και ενεργοποιήσαμε το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αλλά δεν υπήρχε καμία οργανωμένη συνδικαλιστική κίνηση. Δυσκολευτήκαμε ε, να επέμβουμε μέσω του Ταμείου ακριβώς γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό και το αναφέρω. Μιλούμε για τα κοινωνικά δικαιώματα στη φάση εμβάθυνσης της ενιαίας ε, αγοράς ε, και αναγνωρίζουμε τη βαρύτητά τους. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Γιατί τελικά τι έγινε, έκλεισε από την Ιρλανδία και ξανά άνοιξε στην ε, Πολωνία. Δηλαδή ε, στρέφουμε τους ε, εργαζομένους μιας χώρας εναντίον των εργαζομένων άλλων. Η κυρία Άρκιν έχει το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Κύριε καθηγητά, ε, με χαρά διάβασα την έκθεσή σας. Ε, ε, έπιασα τον εαυτό μου να γνέφει καταφατικά όσο διάβαζα τη σελίδα και να σας πω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, αλλά άκουσα τι υπόθηκε στην Ολομέλεια νωρίτερα. Κάποιος περιέγραψε ως σεξι την εκθεσή σας. Ε, ε, φαίνεται λοιπόν ότι άρεσε σε πολλούς ανθρώπους. Ε, όπως σας είπα δεν ήταν δικά μου τα λόγια αυτά. Αλλά εκτιμώ την ανάλυση σας για την κατάσταση, ιδιαίτερα την ανάλυση πριν την κρίση και μετά την κρίση. Και νομίζω ότι πετύχατε ακριβώς το στόχο όταν είπατε ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πια την αγορά. Είναι καλός υπηρέτης αλλά κακός αφέντης. Και πιστεύω ότι πολύ συχνά οι πολίτες πιστεύουν ότι η αγορά έχει γίνει Αφέντη και γι' αυτό δεν έχουν πίστη σε αυτήν. Ε, αναφερθήκατε ε, στο όχι της Γαλλίας και των κάτω χωρών ε, στην Ιρλανδία. Ε, έζησα δύο εκστρατείες για να πετύχουμε ένα ναι στην συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά νομίζω ότι πολύ συχνά ο κόσμος ξεχνάει το όχι της Γαλλίας και των κάτω χωρών. Ε, έχουν αλλάξει οι δομές στο μεταξύ ε, και δεν ζητήθηκε η γνώμη των ανθρώπων. Ε, δεν το καταδικάζω αυτό, αλλά απλά σας περιγράφω τι συνέβη και αυτό είναι συμπτωματικό του γεγονότος ότι ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη το να, να ξαναγυρίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην Ιρλανδία δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το λέω σήμερα, μπορεί ο κόσμος να ε, υπερβάλλει, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων ε, στην Ιρλανδία που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης ε, Λαβάλ και Ρούφος ε, είναι πολύ μεγάλος, διότι θεωρούν ότι αυτό αποτελεί άμεση συνέπεια στις ζωές τους. Ε, και ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει αυτό ήδη εδώ. Δύο παρατηρήσεις ε, θα κάνω και έχω και μετά ε, ερωτήσεις. Μία παρατήρηση. Είπατε και συμφωνώ απόλυτα ότι η πιο ισχυρή εσωτερική αγορά δεν θα επιτευχθεί χωρί ε, τη συνένεση και αναφέρεστε στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πολίτε και τους καταναλωτέ. Ε, και συμφωνώ απόλυτα με ε, αυτό και πιστεύω ότι μια σειρά από τι, συστάσεις σας, ελπίζω μια σειρά από τις συστάσεις σας να υιοθετηθούν και να μα οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά έχω τρει ερωτήσει που θέλω να σα θέσω. μιλήσατε για δημοσιονομική παγίωση. από την Ιρλανδία προέρχομαι. εάν τηρήσουμε τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας μέχρι το 2014, η αριθμητική σημαίνει ότι ε, θα έχουμε πρόβλημα με την οικονομία μας και νομίζω, υποψιάζομαι ότι αυτό είναι αλήθεια και για, κάποιες, και για κάποια άλλη κράτη-μέλη. Όπως και άλλα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει ε, να βρούμε τα σωστά νούμερα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε, θα βλάψουμε μακροπρόθεσμα τις οικονομίες μας, η μακροπρόθεσμη ανεργία θα αυξηθεί ραγδαία θα ήθελα λοιπόν τις απόψεις σας για τη συγκεκριμένη ε, περίπτωση. Η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με τον συντονισμό των φορολογικών συστημάτων. Εάν υπήρχε ε, αίσθηση στην Ιρλανδία ότι θα υπάρξει φορολογική, ε, φορολογικό συντονισμό, τότε δεν νομίζω ότι θα είχαμε πετύχει το ναι στην Λισαβόνα κατά το δεύτερο δημοψήφισμα. Θα ήθελα τη γνώμη σας όσον αφορά την πρόοδο που γίνεται σχετικά με μια κοινή φορολογική βάση για το, τη φορολογία των επιχειρήσεων. Αυτό έχει να κάνει με το πού παράγονται τα προϊόντα, πού πολλούνται, μπορεί ε, να γίνει κάποια δίκαιη κατανομή των ε, φόρων ε, μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα ε, τις παρατηρήσεις σας σχετικά με αυτό. Και τέλος είπατε για την ενιαία αγορά ότι θα πρέπει να την αφήσουμε ανοιχτή, να μην την αφοπλίσουμε όμως και νομίζω ότι ε, είναι πολύ καλός τρόπος περιγραφής του πώς πρέπει να δούμε την παγκόσμια προοπτική. και κάποιοι συνάδελφοι το ανέφεραν. Θα ήθελα πολύ όμως να ακούσω τη, γνώμη σας, τη σκέψη σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρεζίνα Μπάστος και μετά η κυρία Ελίζα Πεθσρέντερ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον καθηγητή Μόντι για τον ενθουσιασμό που δείχνει και την ελπίδα που μας μεταφέρει όταν παρουσιάζει την πολιτική του για την τόνωση της ενιαίας αγοράς, την ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς που θα συμπεριλάβει και τα κοινωνικά μέτρα. Ε, μεσούσης της κρίσης ε, οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινωνική διάσταση όπως σωστά είπατε, αλλά ε, υπάρχουν διάφορα προσκόμματα που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή είτε σε επίπεδο ένωσης είτε σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, έχουμε σοβαρότατα προβλήματα που απορρέουν από την ε, οικονομική ε, και κοινωνική κρίση που οδηγούν σε εθνικό προστατευτισμό. Ορισμένες φορές ακόμη και αιτιολογημένα έχουν εσωστρεφεί στάσεις τα κράτη. Ταυτόχρονα έχουμε την πολιτική 2020 ε, όπου τονίζεται όπως και στη δική σας μελέτη ότι πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση στην Ευρώπη. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, δηλαδή για να ε, εξέλθουμε της ε, κρίσης οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον οικονομικό και στον κοινωνικό τομέα. Βέβαια προς το παρόν υπάρχουν αντίθετα μηνύματα, αντίθετες ενδείξεις ε, ε, που σχετίζονται με την κατάργηση όλων των περιορισμών για την κυκλοφορία των ατόμων, των αγαθών, είτε μιλάμε για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οπότε, θα ήθελα να μας πείτε γιατί δεν σημειώνεται πρόοδος για την αναγνώριση των προσόντων, των επαγγελματικών προσόντων. Για να μπορέσουμε να προαγάγουμε την κυκλοφορία των εργαζομένων. Πώς είναι δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος ενώ υπάρχουν ε, προβλήματα σε εθνικό επίπεδο για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, υπάρχουν ε, διαφορές ε, ως προς τα επαγγελματικά προσόντα ανάμεσα στις βόρειες και στις νότιες χώρες, παραδείγματος χάρη, ένα από τα προβλήματα. Τώρα για το άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης. Έχει μεγάλη πολιτική βαρύτητα τα κράτη-μέλη επιθυμούν την ε, αυτόνομη διαχείριση των ασφαλιστικών συστημάτων τους. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν ε, να οδεύουμε προς μια εναρμόνιση για να προωθήσουμε την ε, κυκλοφορία των εργαζομένων ταυτόχρονα όλοι, ε, όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να συντηρήσουν την ευβιωσιμότητα των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων τους ενώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης. Τέλος, ε, τα δικαιώματα στον τομέα της υγείας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε μία απόπειρα ε, να υπάρξει διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας για να τονώσουμε έτσι την κινητικότητα των ασθενών. Και αυτό σχετίζεται και με την κυκλοφορία των εργαζομένων. Αλλά Ε, Α χρησιμοποιήσω μία ήπια διατύπωση. Δεν απερίφθη το αίτημα, αλλά δεν έγινε δεκτό στο Συμβούλιο. Ε, πώς βλέπετε αυτό το θέμα? Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να συμφιλειωθούν όλα αυτά τα ε, στοιχεία, δηλαδή η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς να συμφιλειωθεί με την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρο. Θα ακούσουμε και την κυρία Σόντε σε αυτό το γύρο ερωτήσεων και μετά πάλι τον ε, κύριο Μόντι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Εμένα θα με ενδιαφέρε να εμβαθύνετε στα δύσκολα ερωτήματα της έκθεσης αυτής. Ένα από τα βασικά δύσκολα ερωτήματα είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινού συμφέροντος, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, και το γεγονός ότι δεν είναι ε, θέμα ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση με τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εμπόδιο ε, στην εσωτερική αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτής όπως ήδη είπα δεν προχωράτε τόσο, είσαστε πολύ πιο επιφυλακτικός και αφήσω ουσιαστικά. Εμένα με ενδιαφέρει ακριβώς αυτό. Στο μέλλον πώς θα είναι τα πράγματα, οι κανόνες εσωτερικής αγοράς θα ισχύουν για ε, κοινωνικές υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος η Κομισιόν θα προσπαθήσει να ρυθμίσει τις υπηρεσίες αυτές με κανόνες της εσωτερικής αγοράς ή θα σεβαστεί αυτόν τον φραγμό που έχει θεσπίσει η συνθήκη της Λισαβόνας και ποια είναι ε, ε, ποια είναι, ποια είναι τα τούβλα αυτού του φραγμού. Ε, δηλαδή, ποιοι είναι οι κανόνες, τι θα πρέπει να γίνει ώστε μία υπηρεσία να μην ε, καλύπτεται από τους κανόνες αντιγραμμιστικότητας αυτούς ε, και τι θα πρέπει να γίνει ώστε να υπάρχει ελευθερία, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στο κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών και όχι στην οικονομική πτυχή. Είναι θέματα που ε, συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες αυτές. Είναι πολύ δύσκολο να ε, αναπτύξουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Ε, υπάρχει... Άκουσα ότι υπάρχει μια πολύ καλή μελέτη του Ιδρύματος του Δουβλίνου σήμερα το απόγευμα ε, που δείχνει ότι θα οδηγηθούμε σε κοινωνικό διχασμό. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό ε, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική πτυχή. Ευχαριστώ. It's very instructive for me to come to this committee. Είναι πολύ χρήσιμο για μένα να βρίσκομαι στην Επιτροπή αυτή, διότι επιτέλους βρίσκω να υπάρχουν θέματα τα οποία γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ή άλλες ε, ή άλλες επιτροπές. Ε, Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, δεν την ακούσαμε. Να απαντήσω με τη σειρά. Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την υπόθεση Dell, και ε, τις τοπικές διαστάσεις. Ε, να σας θυμίσω ότι πέρα από τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα πιστεύω ότι είναι σημαντικό όπως σημειώνεται στην έκθεση αφενός να εισάγουμε μία ρήτρα προϋποθέσεων για τα διαφθορτικά ταμεία, ώστε να ανταμείψουμε τα κράτη-μέλη που ήταν πιο συνεπείς στη μεταφορά των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς στο εθνικό τους δίκαιο. Οι χώρες λοιπόν θα θα επωφελούνται από τη συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά Ε, συμπεριλαμβανομένου του όφελους ε, να ε, λειτουργούν ως τόποι παραγωγής. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ρήτρε για τα διαφθορτικά ταμεία που να ανταμείβουν τα κράτη-μέλη που όχι μόνο υποφελούνται από την εσωτερική αγορά αλλά και που συμβάλλουν σε αυτήν ε, με την γρήγορη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των σχετικών οδηγιών. Ε, ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία ε, είναι η θέσπιση κανόνων που να εμποδίζει την χρήση των διαφορετικών ταμείων για να στηριχθούν οι τόποι παραγωγής επιχειρήσεων. Κυρία Χάρκιν, δεν γνώριζα την δεν γνώρισα ότι μια έκθεση για τη νέα στρατηγική της εσωτερικής αγοράς μπορεί να είναι σεξι, κυρίως ε, επειδή κάτι που πάντα λέω είναι ότι δυστυχώς το θέμα της εσωτερικής αγοράς δεν είναι καθόλου σεξι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντική δυσκολία. Πολλά άλλα θέματα είναι πολύ πιο ελκυστικά από πολιτικής άποψης όπως όλα τα θέματα που συζητάει η Επιτροπή για την κρίση. Η κρίση εξορισμού είναι σεξι, δεν είναι. Το πολιτικό σημείο κλειδί είναι το πώς να μεταμορφώσουμε την ενιαγορά. Είναι, δεν είναι καθόλου σεξι, είναι γκρίζα, γραφειοκρατική, έχει ένα σωρό μειονεκτήματα. Εκτός από το ότι αποτελεί τη βάση του ευρώ ε, για τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αποτελεί δηλαδή τη βάση που ε, σήμερα για καλούς κακούς λόγους είναι πολύ πιο ελκυστικά από πολιτικής πλευράς. Το πρόβλημα είναι λοιπόν πώς να προσελκύσουμε το πολιτικό ενδιαφέρον στον ε, πυλώνα που τα στηρίζει όλα αυτά, δηλαδή την εσωτερική αγορά. Ε, πιο συγκεκριμένα για τα επιμέρους ζητήματα που αναφέρατε. Ναι, η δημοσιονομική ε, παγίωση, όπως είπατε, μπορεί να μας απομακρύνει από την ανάπτυξη. Ωστόσο πιστεύω ότι όταν η κοινή γνώμη και οι αγορές ταράζονται, κλονίζονται από υψηλά ελλείμματα και χρέη, σε κάποιο βαθμό η δημοσιονομική παγίωση μπορεί να και σταθεροποίηση μπορεί να βελτιώσει τις προσδοκίες, το λεγόμενο αποτέλεσμα Ρικάρντο, το οποίο μπορεί ε, να ενεργήσει ε, ως διεύρυνση και όχι ως περιορισμό. Ε, αλλά πιστεύουμε ότι ε, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μπορεί να έχουμε ακριβώς το περιοριστικό αποτέλεσμα και σημαντικό είναι να το αντισταθμίσουμε αυτό ε, με μια δυναμική πολιτική όσον αφορά την προσφορά, ώστε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και την εσωτερική αγορά. Ε, όσον αφορά τον συντονισμό των φορολογικών συστημάτων, ε, στις διαβουλεύσεις που είχα, ε, διαπίστωσα ότι οι επιχειρήσεις είναι πολύ υπέρ αυτού. Φυσικά, πολλά κράτη-μέλη είχαν ιδιαίτερη δυσκολία με το θέμα αυτό. Αναρωτώ ε, εάν έχει επενδυθεί αρκετή πολιτική προσπάθεια στο θέμα αυτό και σε άλλα ζητήματα φορολογικού συντονισμού. Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση είναι πως όχι. Και πιστεύω ότι όταν ξεκινήσει μια πολύ πιο ισχυρή παιδαγωγική και πολιτική δράση, τα κράτη-μέλη θα είναι πολύ πιο ανοιχτά απέναντι στο ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά την ανοιχτή και όχι αφοπλισμένη εσωτερική αγορά, Θέλατε περισσότερες πληροφορίες. Ε, ξέρω ότι ε, ο Επίτροπος Δεκούχτ ε, εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες μόχλευσης που έχουμε. Για παράδειγμα γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν τρελαίνεται για τις διμερείς συμφωνίες με την Νότια Κορέα για άλλους λόγους, αλλά στην συμφωνία αυτή υπάρχει μια ρήτρα όσον αφορά την ε, πειθαρχία στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που ε, αποτελούσε πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μπάστος. Ε, έχετε πολύ βαθιά και άμεση γνώση από τα συγκεκριμένα προβλήματα βλέπω και, τα, και τους φραγμούς στους οποίους έχουν ε, ε, περισσότερες αντιρρήσεις τα κράτη-μέλη όσον αφορά την κινητικότητα, την ε, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και το πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσέγγισης όσον αφορά την καταπολέμηση κάποιων προνομίων που υπάρχουν ή κάποιων χασμάτων που δημιουργούνται. Ε, για παράδειγμα το θέμα των ε, πολιτικών μηχανικών από την Ισπανία ε, στην Πολωνία, διότι είδαμε ότι μετά το τέλος της ανάπτυξης στον οικοδομικό τομέα πολλοί πολιτικοί μηχανικοί δεν έβρισκαν δουλειά στην Ισπανία και ήθελαν να πάνε στην Πολωνία. Υπάρχουν όμως κανόνες που, αν θυμάμαι καλά, σημαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν και γνώση της ε, πολωνικής γλώσσας, που νομίζω ότι είναι ε, αναλογική απέτηση όσον αφορά έναν γιατρό. Δεν είμαι όμως βέβαιος αν αυτό θα πρέπει να ισχύει και για έναν πολιτικό μηχανικό. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε συνδυασμό δράσεις ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως αρχής για τον ανταγωνισμό και δράσεις σε επίπεδο αμοιβαίου ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών. Συμφωνώ όμως, ε, αναφέρατε και το δικαίωμα στην ε, ιατρική περίθαλψη, την κινητικότητα των ασθενών. Αυτά είναι ακαθόδη θέματα. Πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν ε, εάν τα συνδυάσουμε σε ένα πακέτο, διότι κάποια, κάποιες από τις χώρες που προβάλλουν τη μεγαλύτερη αντίσταση στα μέτωπα αυτά, που είναι πιο αντίθετες στο άνοιγμα τους, είναι και οι χώρες που θα ήθελαν να δουν πρόοδο, για παράδειγμα, στον τομέα του φορολογικού συντονισμού. Εάν λοιπόν είναι δυνατόν να φτιάξουμε ένα πακέτο, το οποίο να περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία, διάφορα στοιχεία, μπορεί να είναι δυνατόν να πετύχουμε πρόοδο σε θέματα όπου βλέπουμε πεισματική αντίσταση ε, σε θέματα όταν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Τα πράγματα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνδυαστούν σε ένα πακέτο. Κυρία Σρέτερ ομολογώ ότι η γνώση μου των κοινωνικών ζητημάτων που αναφέρατε είναι περιορισμένη. Σημειώνω ότι είπατε ότι η έκθεσή μου δεν προχωράει αρκετά όσον αφορά ε, τις ε, υπηρεσίες ε, κοινού ενδιαφέροντος. Να σας διαβεβαιώσω όμως ότι στην Επιτροπή πολλοί πιστεύουν ότι η έκθεσή μου ε, προχωρά υπερβολικά σε κάποια θέματα. Και πιο γενικά όσον αφορά την ε, πιο ισχυρή κοινωνική διάσταση, αναρωτιέμαι αν αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί, ε, επιτευχθεί με πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με συντονισμό δηλαδή, ε, ή όπως θα έτεινα εγώ να πιστεύω χωρίς να είμαι ε, εμπειρογνώμονας στις κοινωνικές πολιτικές όπως είστε εσείς, θα έτεινα να πιστέψω ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε κάποια από ε, κάποιες από τις παρενέργειες ε, τη ενιαία αγορά που δυσκολεύουν ε, τις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών να επιδιώξουν τους κοινωνικούς τους στόχους. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ισχύει στο θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού. Εάν δεν τον ελέγξουμε, θα διαβρώσουμε τη φορολογική βάση, θα στρεβλώσουμε την φορολογία υπέρ του κεφαλαίου και κατά της εργασίας και θα δυσκολέψουμε τα κράτη-μέλη στην ε, ε, δημιουργία των δικών τους ε, κοινωνικών πολιτικών για να βοηθήσουν τους χαμένους μέσω των προϋπολογισμών τους. Αυτές οι συνοδευτικές πολιτικές λοιπόν πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές για να υπάρξει περισσότερη ελευθερία όσον αφορά την κοινωνική διάσταση. Δεν θέλω όμως αυτές οι απαντήσεις που έδωσα στην τελευταία σειρά ερωτήσεων να θεωρηθεί ότι είναι πλήρης ε, εις βάθος απαντήσεις. Δεν είναι. Είναι διαστάσεις αυτές όπου ειδικά η Επιτροπή σας θα μπορέσει να συμβάλλει σημαντικά ε, όταν ε, δούμε τις συστάσεις της Επιτροπής που θα ακολουθήσουν την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τις τελευταίες ερωτήσεις, η κυρία Μοχάν και η κυρία Φιγκυρέντο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, καθηγητά. Ε, ε, ε, διάβαζα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ολόκληρη τη μελέτη σας και έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα να σας θέσω. Κατανοώ τον προβληματισμό που μπορεί να έχουμε σε οικονομικό επίπεδο, αλλά στη δική μας επιτροπή ασχολούμαστε με τις επιπτώσεις των οικονομικών επιλογών επί των όρων διαβίωσης ε, των γυναικών και των αντρών. Επιθυμείτε να έχουμε μία ανοιχτή ε, ενιαία αγορά για να αντιμετωπίσουμε το διεθνή ανταγωνισμό. Όμως, όπως είπε και η συγκήτρια, ε, καθήκον μας είναι να μελετούμε τη δράση του Κοινωνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και παρακολουθούμε την πορεία των ευρωπαϊκών εταιριών και των μισθωτών τους που πλήττονται σφόδρα από την κρίση. Ε, έχουμε πολλοί άριθμα και λένε και περισσότερα αιτήματα για βοήθεια μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης για ένα δύο ε, αριθμό μισθωτών. Οι χώρες BRIC ε, ε, λοιπόν αποτελούν τον σημαντικότερο διεθνή ανταγωνισμό. Πώς ακριβώς προτείνεται να έχουμε μια ισορροπημένη ενιαία αγορά. Μιλήσατε για γεωγραφική κινητικότητα. Ε, αλλά δεν έχει ε, τονωθεί επαρκώς ε, ούτε και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και πάντοτε, αντί να λειτουργούμε προληπτικά με τα προγράμματά μας, αντιδρούμε στις εξελίξεις. Και πάλι λοιπόν, μεσούς της κρίσης, πώς να κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε άμεσα αυτή την κρίση και ανάντι να κινηθούμε για να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους εξασφαλίζοντας ε, ε, ταυτόχρονα ε, πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των μισθωτών, αλλά αντιμετωπίζουμε σοβαρότητα τις δυσκολίες, εμοραγεί η ευρωπαϊκή οικονομία, κλείνουν εταιρείε λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού, λόγω του ανταγωνισμού των χωρών BRIC. Ε, και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Η ε, πρόεδρος. Ε, έχει αποχωρήσει η κυρία Φιγκυρέιτο. Νομίζω ότι θα διαπραγματεύεται έξω τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα μιλήσω εγώ αντί για αυτήν λοιπόν. Καθηγητά, από την αρχή της θητείας σας, σας έχω κάνει μια ερώτηση και θα την υποβάλω και πάλι σήμερα. Σημαντική είναι η εσωτερική αγορά για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύτιμη. ναι, όλα αυτά καλά και σωστά, αλλά ε, μέσα στα πλαίσια της ε, μελέτης σας ε, προκύπτει και το εξής πρόβλημα. Ποια, σε τι βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση η ελεύθερη, στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των αγαθών των ανθρώπων. Ε, και όπως ε, κάνατε και αυτό τον παραλληλισμό με την Αμερικανική ε, αγορά, ε, στηρίζεται στην φορολογική εναρμόνιση και τονίζω φορολογική εναρμόνιση και όχι συνεργασία, την δυνατότητα διασυνοριακής πρόσβασης στις υπηρεσίες κτλ. Αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία. Ε, και επίσης μας μιλήσατε για τις συναντήσεις ε, που είχατε με τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, στα πλαίσια της ακρόσης που διοργάνωσε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και εκεί αναφερθήκατε στην δυσκολία εξέβρεση ισορροπίας και συμφιλίωσης ανάμεσα στην ενιαία αγορά και τις εθνικές αγορές. Αλλά τι ισχυριζόμαστε ότι έχουμε την οδηγία για τις ε, υπηρεσίες ε, και ε, πραγματώνουμε την ενιαία αγορά, μα αφού δεν σημειώνεται πρόοδος. Ξέρετε, όλα τα επιμέρους στοιχεία πρέπει να προχωρήσουν εκ παραλίλου. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συνοχή του πακέτου μέτρων που καθίστανται αναγκαία. Πώς απαντάτε λοιπόν στο φορολογικό ζήτημα. Μιλήσατε για τη συγκρότηση μιας ειδικής επιτροπής για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, εγώ ε, ξέρω ότι στο Συμβούλιο υπάρχει αρμόδια ομάδα εργασίας. Τι πρέπει ε, να κάνουμε, που εξετάζει το τι πρέπει να κάνουμε για να εφαρμοστούν οι προτάσεις σας. Εσείς έχετε ολοκληρώσει το έργο σας, αλλά φαντάζομαι σας ενδιαφέρει να ξέρετε αν υλοποιούνται, αν εφαρμόζονται, αν αξιοποιούνται οι προτάσεις σας από τα θεσμικά όργανα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Μωρά με εικαστικό τρόπο περιέγραψε την διόγκωση των προβλημάτων λόγω του ανταγωνισμού των χωρών BRIC και άλλων. Νομίζω ότι από μόνη της η ενιαία αγορά δεν θα μας δώσει την απάντηση Βλέπουμε ότι ε, με σαφήνεια ότι ο κατακαιρματισμός ενιαίας αγοράς και η αύξηση του εθνικού προστατευτισμού σίγουρα επίσης δεν συνιστούν απάντηση στα προβλήματά μας. Ορισμένε φορέ ε, τίθεται να αμφιβόλω το ευρύτερο όραμα ε, τη Ευρώπη ε, λόγω των συρρυκνούμενων δημοσιονομικών πόρων, των οικονομικών προοπτικών. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον το Κοινωνικό Ταμείο Αλληλεγγύης. Αλλά σίγουρα δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές προκλήσεις ε, στα, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα επανέλθω σε αυτό το πακέτο ε, μέτρων που πρότεινα και την ε, παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων, αυτό που με ρωτήσατε εσείς Πρόεδρε. Ε, προχωράει η φιλελευθερωποίηση της αγοράς, ε, αλλά ταυτόχρονα μένουμε μόνο στα υπεσχημένα ε, όταν ε, πρόκειται για την φορολογική εναρμόνιση. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι πρέπει στα δύο μέτωπα ε, ταυτόχρονα να σημειωθεί πρόοδος. Γιατί αλλιώς ε, δεν υπάρχει ελπίδα για την αγορά. Un Στις 20 Ιουλίου με έχει προσκαλέσει ο πρόεδρος Μπαρόζο σε μια συνεδρία του Σώματο των Επιτρόπων για να ε, συνομιλήσω με τους συναρμόδιου επιτρόπους και να ε, παρακολουθήσω την συνέχεια που εδόθη στη μελέτη μου. Ξέρετε ότι υπάρχει και η, έκθεση, η ελληνική έκθεση πρωτοβουλία στην Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου dans les différentes ε, και ε, κάθε επίτροπος ε, και κάθε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Πρέπει να παρακολουθήσουμε λοιπόν τα επιμέρους στοιχεία του πακέτου αλλά και σφαιρικά το πακέτο. Γιατί πρέπει εκ παραλλήλου να σημειωθεί πρόοδο σε όλους αυτούς τους επιμέρους τομείς. και η συμβολή ε, του Πρόεδρου της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχει ιδιαίτερη σημασία διότι χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική ε, που σχετίζεται με το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων, ανταγωνιστικότητας, οικονομικών υποθέσεων, και άρα χρειάζεται πολιτική ηγεσία. Ο μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να επιληφθεί της υπόθεσης Φέρικα γιατί ε, ήδη ασχολείται με την οικονομική διακυβέρνηση και αυτό πρέπει, το κοινωνικό κομμάτι πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διακυβέρνησης και στα τρία ε, θεσμικά όργανα νομίζω χρειαζόμαστε πιο ολιστική προσέγγιση, σφαιρικότερη προσέγγιση. Πάντως ε, η ρόλη είναι ε, ξεκάθαρη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, και φυσικά είναι θεματοφύλακας των συνθήκων. Ως προς την νομοθετική διαδικασία για τα ζητήματα ενίας αγοράς, πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ακολουθηθεί ε, σπευσμένη διαδικασία και από το Κοινοβούλιο και από ε, το Συμβούλιο, όπως έγινε και το 85, έτσι, μετά την ε, Λευκή Βίβλιο Ντελόρ. για να υπάρξει ε, ενιαίο κοινό όραμα και να επισπευστεί η πρόοδος. Θα παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς ε, την πρόοδο των εργασιών σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την ε, σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Ε, ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα. Ε, μήπως έπρεπε να είχαμε καλείς και νωρίτερα συνειδητοποιώ τώρα που σας άκουσα. Τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά πότε. Ε, πρέπει να κινητοποιηθούμε για το πακέτο μέτρων ούτω ώστε να στεφθεί με επιτυχία το όλο εγχείρημα σε όλες τις διαστάσεις του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία συνάδελφοι. Θα επανέλθουμε τώρα στην κανονική μας ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ να είστε συνοπτικοί για να προλάβουμε. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ και ο κύριος Άνταμ ε, Κόσα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις ε, από τη Σκιώδη. Για μας το θέμα της οδηγίας πλαίσιο είναι αρκετά σημαντικό διότι προσπαθούμε να καθορίσουμε ε, κάποια πρότυπα και κάποιες κοινέ απόψεις για το πώς φτάσαμε σε αυτή την κοινή άποψη για το ελάχιστο εισόδημα έχει σημασία για την πρόσβαση, για τη συμμετοχή και φυσικά για την καταπολέμηση της ένδυας, για να μπορεί κάποιος να ζει με αξιοπρέπεια. Μας ενδιαφέρει πολύ λοιπόν η τροπολογία 133 και η συνέχεια που θα έχει. Ε, από αυτήν προέγυψε ο συμβιβασμός M. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είμαστε με αυτό το συμβιβασμό, αλλά τέλος πάντων. Εν είδη εξήγησης, όταν θα το ψηφίσουμε αυτό αύριο, υπάρχουν κάποιε τροπολογίε από σκανδιναβού συναδέλφου που μα δημιουργούν προβλήματα. Διότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ελάχιστου εισοδήματο και ελάχιστου μισθού. Και παρά το γεγονό εκτιμούμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε αρκετέ κράτη-μήλε, στι ε, συλλογικέ ε, συμφωνίε μισθών, δεν έχουμε το ίδιο στοιχείο στο ελάχιστο εισόδημα όταν κάποιος είναι άνεργος και συμμετέχει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε λοιπόν κάποιες επιφυλάξεις με τις τροπολογίες αυτές. Δεν είμαστε ακριβώς αντίθετοι, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι λένε ακριβώς αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε να πούμε εμείς αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο Άνταμ Κώσας και μετά ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν προφέρατε σωστά το όνομά μου και δεν κατάλαβα τι έπρεπε να παρέμβω εγώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. διότι ασχολήθηκε με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. παρουσίασα κάποιες τροπολογίες, κυρίως για τα άτομα τα οποία είναι βέλατα σε διάφορα επίπεδα. Καταρχάς αναφέρομαι στα άτομα με αναπηρίες προφανώς, διότι τα άτομα με αναπηρία είναι αυτά τα οποία είναι περισσότερο εκτεθισμένα σε κινδύνους, ε, κυρίως κινδύνους ένδυας. Και εδώ έχουμε και το θέμα της ε, γύρανσης, διότι θεωρώ ότι η τρίτη ηλικία και η αναπηρία είναι αλληλένδετα στο σημερινό κόσμο. Όσον αφορά στις συμβιβαστικέ τροπολογίες, ε, δέχομαι ε, με πολύ ευνοϊκό τρόπο το γεγονός ότι βρήκαμε κάποιες ε, θετικές λύσεις υπό την έννοια ότι οι ομάδες στόχος έχουν μείνει μέχρι το τέλος στο συμβιβασμό. Τώρα, για μια συγκεκριμένη συμβιβαστική τροπολογία θα ήθελα να επισημάνω ότι ίσως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη την άρση των ε, εμποδίων για την πρόσβαση στις κοινωνικές ε, ε, υπηρεσίες. Αναφέρομαι στο συμβιβασμό K για τις δημόσιες υπηρεσίες. Επισημαίνονται εδώ οι δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται και εκχωρούνται από το κράτος ή από τις τοπικές αρχές. Και για αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να διαγράψουμε να, να άρουμε συγγνώμη, και τα φυσικά προσκόμματα αλλά και τα εμπόδια στην επικοινωνία. Επίσης διαπίστωσα ότι υπάρχει μια κάποια δυσαρέσκεια ω προ το γεγονό ότι για αυτή τη συμβαστική τροπολογία διαγράφηκε το βασικό σημείο, δηλαδή ότι μιλάμε για δημόσιε υπηρεσίες. Ολοκληρώνοντα, να πω ότι ελπίζω ότι όλε οι συμβαστικέ τροπολογίε θα γίνουν δεκτέ και είμαι περίεργος να δω σε τι νέες λήξεις θα καταλήξουμε ε, και λόγω της σημερινή συζήτησης. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε όμως και περαιτέρω συζητήσεις και διευκρινήσεις επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ε, ε, Συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ να είστε πιο σύντομοι, γιατί δεν θα προλάβουμε. Ο κύριος Κρίστενσεν και μετά ο κύριος Κονφεράτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε με τη σημαντική αυτή έκθεση. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος μαζί με τους συναδέρφους μου από την Φιλανδία, ε, Γιακονσάρη και Λούντβιξον από τη Σουηδία. Έχουμε υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες. 67, 110, 144. Οι τρεις αυτές τροπολογίες συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικές E, ε, K και M ε, και έχουν γλωσσικό στόχο. Η γαλλική μετάφραση θα πρέπει να είναι η ίδια και σωστή ε, για Μάλλον η ε, ε, γαλλική μετάφραση των συμβαστικών ε, τροπολογιών είναι σωστή, αλλά στα αγγλικά υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες, ιδιαίτερα στις τροπολογίες I και K. Μία μικρή διόρθωση. Μαζί με τους συναδέλφους μου αυτούς έχω υποβάλει τροπολογία υπαριθμών 78, όπου προτείνουμε να διαγράψουμε το δεύτερο μέρος της πρότασης. Επειδή αυτό δεν έχει γίνει στη συμβιβαστική τροπολογία, θα ήθελα να αφαιρεθεί η τροπολογία 78 από το συμβιβασμό. Δεν έχουμε όμως πρόβλημα με τη συμβαστική τροπολογία, απλά αποσύρουμε την τροπολογία 78. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτη και μετά η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω δύο πράγματα πολύ σύντομα. Καταρχάς νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες παρεξηγήσεις λόγω μετάφρασης. Είμαστε στο τέλος μιας πορείας και υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ερμηνεία και αυτό δεν είναι καθησυχαστικό. Μιλάμε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όχι για τον ελάχιστο εγγυημένο μισθό. Ο μισθός είναι καρπός της εργασίας κάποιου είναι η πληρωμή για τη δραστηριότητά του. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο είναι πολύ σαφώς καθορισμένο και ε, είναι ε, πολύ καλά ε, περασμένο στην νομοθεσία. Ενώ η ένδυα είναι πολύ πιο βαριά για ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι. Υπάρχουν μεν φτωχοί εργαζόμενοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι και είναι φτωχοί ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μια επαγγελματική δραστηριότητα και δεν υπάρχει εισόδημα. Θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό, διότι η ιδέα του ελάχιστο κειμένου μισθού είναι, ναι μεν μια πολύ καλή ιδέα, αλλά είναι μια παλιά ιδέα. Τώρα θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες συνιστώσεις ε, οι οποίες μας οδηγούν στο σύνολό τους ε, στο εισόδημα και πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη δεν τις έχουν. Πέραν αυτού, νομίζω ότι τα όσα έκανα η κυρία Φιγκερέιδο με τους κοιόδης εισογητής είναι πολύτιμα. Όλα ε, περιστρέφονται γύρω από τη συμβαστική τροπολογία M. Και το ερώτημα εκεί είναι να έχει κανείς ή να μην έχει μια ευρωπαϊκή οδηγία επί του θέματος. Μου φαίνεται ότι η λύση στην οποία καταλήξαμε είναι πολύ λογική, διότι κυριαρχεί η χρήση της οδηγίας, αλλά δεσμεύεται με την αναγνώριση των διαφορών που υπάρχουν και που κατά πάσα πιθανότητα κυρίως, ε, ε, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους, θα παραμείνουν στα κράτη-μέλη. Εγώ εκτίμησα ιδιαίτερα αυτή την προσπάθεια, είχαν παρουσιάσει κάποιες τροπολογίες που, την, που ζητούσαν την οδηγία. Τελεία. Η διευκρίνηση τώρα αυτών των στοιχείων ευελιξίας που αναγνωρίζουν τις ε, διαφορές μεταξύ των χωρών και αναγνωρίζουν ε, και το γεγονός ότι υπάρχει μια μακρά ιστορία πίσω από κάθε κράτος μέλος τις οποίες δεν μπορούμε να συζητήσουμε και που δεν μπορούμε να επιλύσουμε σε ένα κείμενο ε, καταδεικνύουν ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια και την εκτίμησα ιδιαίτερα. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με το κείμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα διαφορετικά στοιχεία, ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει όχι μόνο την απόψή του, αλλά και όλα όσα προκύπτουν από ε, τα όσα συνέβησαν ε, δεκαετίες και δεκαετίες ολόκληρες για τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται το εισόδημα. Ε, η κυρία Ράπτη αποχώρησε δυστυχώς. Η κυρία Μωράν λοιπόν και η κυρία Γκονζιλό παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι. Κυρία Μωρά, Εν συντομία, ε, μιλέψαμε τον Πασκάλ Γκρουνιέ που υπέβαλε την τροπολογία 132 Στα πλαίσια της ε, καταπολέμησης της φτώχειας ε, λαμβάνουν ε, μέτρα τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες απεφεύγοντας την υπερχρέωση. Το πρόβλημα αυτό θέλουμε να τονιστεί όλος ιδιαίτερος μέσα στην έκθεση. Ε, γιατί θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσει στις τράπεζες, γιατί αυτές ευθύνονται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ε, ευχαριστούμε, η κυρία Γκρούσλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να σας καθησυχάσω, δεν είμαι ταραχμένη, διότι με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγεία μου δεν μπορώ να ταράζομαι. Καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Φιγκερέιδο, ε, για τη δουλειά που έκανε. Υπάρχουν όμως τρία σημαντικά σημεία τα οποία έχει αναφέρει το ΕΛΚ και θα ήθελα να τα συνοψίσω εδώ. Πρώτον, η οδηγία πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα, με την οποία διαφωνούμε, θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, επομένως βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Είμαστε ε, πιο πολύ υπέρ ε, κοινωνικών παροχών, ε, οι οποίες αναφέρονται στη σύσταση του Συμβουλίου, την 924421, η οποία καθορίζει κάποια κοινά κριτήρια για τα κοινωνικά συστήματα. Δεν θα θέλαμε μία οδηγία η οποία να είναι τόσο δεσμευτική, συνεπώς. Δεύτερον, Συμβαστική τροπολογία και η τροπολογία 104. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Κος ε, για το θέμα της πρόσβασης χωρίς ε, φυσικούς φραγμαίους ε, και χωρίς προβλήματα στην επικοινωνία. Αλλά το θέμα της στέγασης, housing, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτή την τροπολογία. Και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο. Επομένως δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή και γιατί αναφερόμαστε πολλές φορές ε, στα θέματα της στέγασης ε, σε πολλά άλλα νομοθετικά κείμενα. Τρίτο σημείο, συμβιβαστική τροπολογία ε ή τροπολογία υπαριθμών 33. Ζητούμε επειδή δεν συμφωνούμε με την ε, συμπερίληψη του όρου λαθρέως, ε, καλύτερα να μιλάμε για μετανάστες και να μην κάνουμε διάκριση μεταξύ λαθρομεταναστών και μεταναστών. Και ο άλλος όρος ε, για τις εθνικές μειονότητες, μεταξύ των οποίων και η Ρωμά, το να αναφέρουμε απλώς μία μειονότητα είναι διάκριση έναντι των άλλων μειονοτήτων. Επομένως, ε, θα θέλαμε να παραμείνει μόνο ο όρος ε, οι εθνικές μειονότητες. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, παρότι δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αληθεύει ότι είναι δύσκολο να είμαι σύντομη δίνοντας τι απαντήσεις, διότι παρόλη τη σκληρή δουλειά όλων μας και να ευχαριστήσω εδώ παρεμπιπτόντας όλους τους συνεργάτες μου, παρόλα αυτά υπολείπονται δυσκολίες μέσα σε συμβαστικές τροπολογίες. Κάποιες δύσκολα μπορούμε να τις ρυθμίσουμε. Όπως είπα, ε, για την τροπολογία ε, παραδείγματο χάρη, το θέμα των ε, μεταναστών και των μενοτήτων, Μπορώ να δεχτώ το αίτημά σας, νομίζω θα γίνει δεκτό από όλους. Είχαμε ήδη ζητήσει μάλιστα από τη γραμματεία να το λάβει υπόψη. Για το θέμα της στέγης, ε, το ΕΛΚ πρότεινε δύο διαφορετικές ε, θέσεις. Εμείς θα μείνουμε στην ε, τωρινή εκδοχή του κειμένου, διότι δεν υποχρεώνει κανέναν αυτή η εκδοχή. να μεριμνά ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα σπίτια για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Αλλά προβλέπεται αντίθετα να υπάρχουν σπίτια με πρόσβαση για τα άτομα ε, με αναπηρίες. Αυτή είναι η θέση και του ΟΗΕ και σε, άλλα, σε άλλες εκθέσεις του Κοινοβουλίου αυτή τη θέση είχαμε επιλέξει και η διατομιακή ομάδα εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία την ίδια θέση έχει. Είναι η αρχή που υπάρχει στην ε, σύμβαση του ΟΗΕ. Ε, και μην ξεχνάτε ότι ε, υπάρχει διχογνωμία ακόμη και μέσα στο ΕΛΚ. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει ε, θέλω να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στο ελάχιστο εισόδημα και τον ελάχιστο μισθό. Μα εδώ ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με το ελάχιστο εισόδημα. Δηλαδή μη ανταποδοτικό σύστημα. Άλλο πράγμα είναι ο ελάχιστος μισθός. Ίσοδυναμή με τις αποδοχές. Το ελάχιστο εισόδημα είναι μη ανταποδοτικό σύστημα. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει τα προστοζήν και χρειάζεται βοήθεια. Του εξασφαλίζουμε αξιοπρεπή σε συνθήκες ζωής. Περί αυτού ο λόγος εδώ και τίποτε άλλο. έχουμε κριτήρια, κανόνες, που, όρους που επιτρέπουν μια ελάχιστη διαβίωση ε, για τους απόρους. Τώρα, ε, συζητούμε εδώ κάτι που απασχολεί το Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Ένα ε, κομμάτι ένα τμήμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχου, έχει λάβει υπόψη αυτό το παράγοντο, αλλά όχι όλα. Και τώρα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ε, λόγω της κρίσης. Μιλώ για ε, τα σημαντικότερα στοιχεία της ε, στρατηγικής ε, καταπολέμησης της φτώχειας και κυρίως για το ακαμφόδες αυτό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εδώ δύο-τρεις ιδέες γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν την χάνουν γενικής αποδοχής σε αυτήν την τροπολογία θα μπορούσαμε να ε, προσθέσουμε μια προφορική τροπολογία όπως αυτή που ε, εισηγήθηκε η κυρία Λίνε ούτως ώστε να μην λέμε πια οδηγία πλαίσιο και να πούμε Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Αντί για Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο να πούμε Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Και ξέρω ότι υπάρχει και μία χωριστή τροπολογία υπαριθμών 88 όπου ζητείται οδηγία, έγκριση οδηγίας πλαίσιο. Θα έλεγα με την ιδιότητα της εισηγήτριας ότι λαμβάνοντας υπόψη αυτή την τροπολογία 88 που μιλάμε για οδηγία πλαίσιο ε, που θα ψηφιστεί ξεχωριστά επειδή είναι ξεχωριστή τροπολογία μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την αναφορά. Δυσκολεύεται η συνάδελφος Λίν ε, να δεχτεί αυτή την συμβαστική πρόταση. θέλει να μιλήσουμε μόνο για ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα οδηγεί σε σχέδιο δράσης, το οποίο ή μάλλον θα υπάρχει ε, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να συνοδεύεται η εθνική πρακτική στον τομέα του του εισοδήματος και μετά συνεχίζουμε εθνικές πρακτικές, συλλογικές συμβάσεις όπως έχει το κείμενο. Θα ε, διαγράψουμε λοιπόν την ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο και θα μιλήσουμε για Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Τώρα, στην τροπολογία 88 δεν αλλάζει τίποτα. Θα παραμείνει η αναφορά στην ε, Οδηγία Πλαίσιο, Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σε πλαίσιο. Άρα θα υπερψηφίσω εγώ προσωπικά την ε, τροπολογία 88. Ε, Είναι μια δυνατότητα που τίθεται επιτάπητος, αλλά Πραγματικά θα ήθελα να γνωρίζω πώς τοποθετούνται οι λοιπές πολιτικές ομάδες, οι φιλελεύθεροι ε, ε, και το ΕΛΚ θα υπερψηφίσουν το σύνολο των συμβαστικών τροπολογιών. Αναρωτιέμαι. Για να επιτύχει αυτό το τελικό, αυτή η τελική απόπειρα, Και ξαναλέω, όσοι συμφωνούν μαζί μου και υπερασπίζονται αυτή την ιδέα τη οδηγία πλαίσιο, α υπερψηφίσουν την τροπολογία 88. Ε, πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα ήθελα ε, να μας δώσετε λίγα λεπτά, ούτω ώστε να τοποθετηθούν εντάχει οι σκιώδεις για αυτό το θέμα. Ε, δεν έχω πρόβλημα ε, να ικανοποιήσω το αίτημά σας, ε, αλλά ναι ή όχι. Καταφατικά αρνητικά θα απαντήσετε και τίποτα παραπάνω, γιατί έχουμε άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Κυρία Ροντζούλη. Όχι, ε, έτοιμη είμαι. Για μας, να τα πω ιταλικά που είναι πιο εύκολο. δεν μας κάνει. Διότι δεν είναι μόνο η τροπολογία 88 το πρόβλημα, Έχουμε και άλλες ε, τροπολογίες στις οποίες αναφερόμαστε στην οδηγία. Ο όρος πρωτοβουλία μας αρκεί, αλλά ή θα το περάσετε σε όλα ή εμένουμε στη θέση μας. Euh, Αν κατάλαβα καλά κυρία Ροντζούλη, δέχεστε τη συμβαστική τροπολογία M με την ε, τροποποίηση που προτείνει η συγγήτρια. τροποποιημένη. Μα σα ρωτάμε αν δέχεστε την ε, συμβαστική τροπολογία M βάσει τη τροποποίησεις που προτείνει η συγγήτρια. Ε, και ε, ακούσατε ότι δεν τροποποιούνται άλλε τροπολογίε για να μπορεί κάποιο να καταψηφίσει την ιδέα. Εσείς δέχεστε την τροποποιημένη τροπολογία, δηλαδή να μιλήσουμε για ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και όχι για την οδηγία πλαίσιο. Αν ε, δεν υπάρχει πρόβλημα, επιφυλάσσομαι, θα διαβιβάσω στην εισηγήτρια αργότερα την απόφασή μα. Όταν θα έχουμε το κείμενο, έτσι, πιο πολύ για να έχουμε το κείμενο. Το έχετε το κείμενο, λέει η Πρόεδρος. Όχι, το τροποποιημένο κείμενο δεν το έχω, λέει η κυρία Ροντσούλη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα ε, η μόνη αλλαγή που γίνεται είναι ότι βγάζουμε την ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο, το διαγράφουμε αυτό, και ανταυτού γράφουμε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Αντικαταστούμε μόνο αυτόν τον όρο. Ωραία, εντάξει, αν μείνει έτσι η τροποποίηση. Ο κ. Φεντερίκ Νταρντάν δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Η κυρία η κυρία Λίν δεν είναι εδώ, λέει η πρόεδρος, αλλά είναι δίπλα τη η κυρία Λίν. Είχατε φύγει με του επισκέπτε σα και νόμιζα ότι δεν είχατε επιστρέψει στην αίθουσα. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εδώ είμαι και θα μπορούσα να δεχτώ να αφαιρέσουμε την οδηγία πλαίσιο και να λέμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να οδηγεί σε σχέδιο δράση, ε, το οποίο θα συνοδεύει την εφαρμογή τη ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το ελάχιστο εισόδημα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι αφαιρούμε το, την οδηγία πλαίσιο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά και προσθέτουμε έτσι πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσα να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Κυρία Λαμπέρ, συμφωνείτε. Είναι το ότι συμφωνείτε με τη γλώσσα του σώματος. Η πράσινη δεν είναι κανείς ε, που να ζητάει το λόγο από τους ε, πρασίνους. φανταζούμε. δεν υπάρχουν ε, δυσκολίες. Πολύ ωραία. Τελειώνει και αυτό το σημείο. Αύριο ψηφίζουμε. Σας ευχαριστώ όλους γιατί συνεργαστήκατε για να βρεθεί μια κοινή λύση και τώρα με μεγάλη καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μπορέιρα πρέπει να του κλέψουμε ένα τέταρτο ένα τέταρτο για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο γιατί είναι σημαντικό. Κυρία Μωρά, έχετε το λόγο για την εξέταση των τροπολογιών. Δεν τις έχουμε ακόμα τις συμβαστικές τροπολογίες, αν δεν κάνω λάθος. Τι είπατε, Πρόεδρε, ότι δεν έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κερδίσω λίγο από το χαμένο χρόνο. Υπάρχει ένα λαθάκι. Στην τροπολογία 53 του κυρίου Έντελ για την παράγραφο 12 του σχεδίου και όχι της παραγράφου 11, 12 είναι το σωστό, γιατί αλλάζουν λίγο τα πράγματα στη σειρά των ε, ψηφοφοριών και ήθελα να σας ενημερώσω όλους για αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο ε, εκπονήθηκε πριν ε, από ε, την ανακατονομή στο Δήμο της σχετική ακρόαση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και πριν από τη σχετική συνεδρία της Ομάδας Προϋπολογισμών και πριν από την αποστολή στην Ιρλανδία για όλους αυτούς τους λόγους Δέκα τροπολογίε συνυπεγράφησαν από τα μέλη της αντιπροσωπείας του κλιμακίου που μετέβη στην Ιρλανδία. Έχουν προσυπογράψει λοιπόν τα μέλη του κλιμακίου που εκπροσωπούσαν πέντε πολιτικές ομάδες αυτές τις δέκα τροπολογίες. Ε, συμβαστικές τροπολογίες δεν υπάρχουν γιατί συνεργαστήκαμε τόσο πολύ που ε, τελικά έχουμε συμφωνήσει επί κάποιων αξώνων. Ε, Όλοι επιθυμούμε ενισχυμένο κοινωνικό διάλογο προς ε, όφελος των μισθωτών, μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών και των ερετών εκπροσώπων σε όλα τα επίπεδα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ε, προστατεύοντας ε, το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης. σε όλες τις διαδοχικές αναθεωρήσεις επιθυμήσαμε να ισχύει μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για τη χρήση των πόρων του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η χρησιμότητά του έγκυται στην ευελιξία των μηχανισμών του. Ήθελα να σταθώ λίγο σε κάποιες λίγο πιο περίπλοκες τροπολογίες, ε, ε, των οποίων καλό θα ήταν να προβληματιστούμε συλλογικά. Ε, τροπολογία 10 της κυρίας Κορνέλισεν ήταν στην αποστολή στην Ιρλανδία, δεν ξέρω αν είναι εδώ, εδώ είναι. Αυτή λοιπόν η τροπολογία 10 ζητά από την Επιτροπή ε, ζητά να μεταθέσει την προθεσμία από τις 24 τους 36 μήνες για την υλοποίηση και με την εμβάνθηση που κάναμε για τη χρήση του Ταμείου Προσαρμογής στην ε, ε, Παγκοσμιοποίηση και του Κοινωνικού Ταμείου διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια πολιτική όπως και για το εκτε Προβλέπονται ε, παρεμβάσεις ε, αφενός ε, διαρθρωτικές και αφετέρου ad hoc όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Τώρα, ε, τροπολογία 15 του κυρίου Νταρντά. Σε αυτήν την τροπολογία ο στόχος είναι να ενταχθούν και οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και είναι πολύ καλύτερη η σύνταξη που προτείνεται. Πολλά και αναφερόμαστε στις τροπολογίες μας ε, στην συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και είδατε τι έγινε με την ΤΕΛ, έτσι, στην Ιρλανδία, γιατί δεν υπήρχαν αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι. Θα ζητήσω κατά τμήματα ψηφοφορία για το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας 15, αν επιθυμείτε να τη διατηρήσετε ακέραιη. Εκεί που μιλάμε για, την, ε, για το ρόλο τους στον τομέα της ζήτησης. Μα σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για εθνική ζήτηση και τίποτε άλλο. Άρα μπορεί να υπάρξει πρώτερη διαβούλευση αλλά ε, υπό την αυστηρή έννοια του όρου δεν έχουν αναγνωρισμένο ρόλο ε, σε αυτό το θέμα η κοινωνική εταιρεία. Είναι ε, κρατικό το ζήτημα. Στην τροπολογία 22, κυρία Ρίαμεν Ρόιτεν, ε, ναι, ε, τα ταχεία επέμβαση του Παγκοσμίου Ταμείου Αλληλεγγύης όταν υπάρχει σοβαρή απειλή μαζικής απόλυσης. Μα δεν μπορούμε όταν υπάρχει απειλή να ζητήσουμε να παρέμβει το Ταμείο. Πρέπει να υπάρχει ε, υπαρκτή, υπαρκτό πρόβλημα μαζικής απόλυσης. Για ε, τις 35 και 43. Μάλλον είναι θέμα μετάφρασης, αλλά θα το πω παρόλα αυτά. Ε, λέει στη γαλλική μετάφραση και στην ελληνική εξάλλου καλές σε εισαγωγικά θέσεις απασχόλησης. Στην ισπανική μετάφραση λέμε ποιοτικέ. Ε, και ε, στη γερμανική λέμε επισφαλής. Ε, πώς θα ψηφίσουμε, δεν είναι εύκολο. Θέλω να ξέρω περί τίνος πρόκειται. Γιατί με όλες αυτές τις διαφορετικές γλωσσικές εκδοχές δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Δεν ξέρω και αν είναι και εύστοχη η τροπολογία. Ας μου πείτε αν πρόκειται για επισφαλή ή για ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης για να καταλάβω. Le, euh, 18. Τροπολογία 48 τώρα. Μπορούμε να ζητήσουμε κατά τμήματα ψηφοφορία για το τελευταίο τμήμα αυτής τη τροπολογία. Περί τίνο πρόκειται. Ένα πρόβλημα και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό. Πρόκειται για μη υπηκός ε, κρατών μελών που όμως είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το ΦΕΜ. Και λέμε στο δεύτερο τμήμα ακόμη και αν διαμένουν σε μια άλλη χώρα. Ειδικότερα εάν αφορά ένα άλλο κράτος μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τι, υπονοούμε εδώ πως μπορεί να ε, υλοποιηθεί το ΦΕΜ ε, για μισθωτούς που δεν είναι πολίτες της Ένωσης. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί βλέπουμε ότι ζητείται η παρέμβαση του ΦΕΜ σε εθνικό επίπεδο ε, για ε, εργαζομένους ε, που μένουν σε αυτή τη χώρα. Αλλά εδώ δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε Πολωνούς που δούλευαν στην Ιρλανδία και επιστρέφουν στην Πολωνία άλλο αυτό και άλλο το να έχουμε ε, επικός τρίτων χωρών και αυτό δεν συνάδει με τις ε, καθηγητήριες γραμμές ε, της δράσης του ΦΕΜΕ. Μου ζητήσατε να είμαι σύντομη πρόεδρε και έβαλα τα δυνατά μου. Κυρία Αρκέν και μετά η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την ε, κυρία Μωρίν για την εξαιρετική της ε, έκθεση και την ε, καλή συνεργασία. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες είναι παρόμοιες με αυτές της κυρίας Μωρίν, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Η τροπολογία 5 της κυρίας Κορνέλησεν, ο τρόπος διατύπωσης δεν είναι πολύ καλός, μάλλον είναι γλωσσικό το θέμα, να το κοιτάξουν οι υπηρεσίες παρακαλώ. Το επόμενο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η δική σας ε, τροπολογία, κυρία Πρόεδρε, η παριθμών 12. Συμφωνώ να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά εσείς λέτε ότι οι κοινωνικοί εταίροι βοηθούν να διατυπώσουν τα προγράμματα μετατροπής. Ε, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη τι σημαίνει αυτό. Η κυρία Μωρέν είπε ότι είναι ε, εθνικό ζήτημα, αλλά οποιαδήποτε τροπολογία καλή σε πλήρη συμμετοχή, όχι συνεργασία, πλήρη συμμετοχή των ε, κοινωνικών εταίρων ε, θα έχει την υποστήριξή μου. Τροπολογία 13, την βρήκα λίγο περίεργη, λέει... Ε, αναφέρεται στον κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ε, επιχειρηματίες. Ε, αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω. Συμφωνώ με την κυρία Μωρέν για, το σημείο, για την τροπολογία 15 να έχουμε χωριστή ε, ψηφοφορία. Όσον αφορά την τροπολογία 17 εξετάζουμε την εθνική νομοθεσία στο σημείο αυτό και ένα ερωτηματικό, μάλλον δεν μπορώ να στηρίξω την τροπολογία 19, τουλάχιστον όχι στο σύνολό τη. Όσον αφορά την τροπολογία 23, έχω μία ερώτηση. Λέει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει την συμμετοχή όλων των ε, εργαζομένων ε, που έχουν ε, απολυθεί λόγω, κάποιον λόγω ενός γεγονότος. Νόμιζα ότι το Ταμείο το επιτρέπει αυτό, πως μπορεί η Κομισιόν να μας πει αν ισχύει αυτό ή όχι. Επίσης, η τροπολογία της κυρίας Κορνέλης εν υπαριθμών 24. Αναφέρεται στο να ξεπεράσουμε το διαχωρισμό ανάμεσα στους άνεργους εργάτες μιας κατηγορίας και τους υπόλοιπους. Το EGF είναι κάπως ε, ειδική περίπτωση. Δεν είμαι βέβαια ότι μπορούμε, ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε ε, τον διαχωρισμό αυτό. Ε, επίσης, τροπολογία 31. Και εδώ έχουμε ζητήσει ξεχωριστή χωριστή ψηφοφορία δεν είμαι βέβαια αν μπορούμε να χειριστούμε το θέμα αυτό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Ε, υπάρχει και το θέμα των καλών θέσεων εργασίας, ε, μπορεί και αυτό να είναι θέμα μετάφρασης ε, και υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε για την παράγραφο 7. Σημειώνω ότι η συγγήτρια της στηρίζει αυτέ και εγώ θα στηρίζω τι περισσότερε από αυτές. Φοβάμαι όμω ότι αν υιοθετηθούν όλες θα καταλήξουμε σε ένα πολύ μακρύ κατάλογο με καλέ θέσει απασχόληση, πράσινε θέσει απασχόληση, βιώσιμε θέσει απασχόληση. Ε, δεν είμαι σίγουρη ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τροπολογία 40. Δεν μπορώ να τη στηρίξω, διότι λέει ε, ότι η ανεργία οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση. οι περιπτώσει απολύσεων οι οποίε προκαλούνται από την ε, παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι πολλοί από εμά έχουμε σοβαρέ συντηρήσει για το θέμα αυτό. Ε, τροπολογία 44, το τελευταίο κομμάτι σε έναν διαχρονικά σταθερό τομέα. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν. Μήπω μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμε θέσει απασχόληση, αυτό θα είναι καλύτερο. Τέλο, ε, και νομίζω θα κλείσω η τροπολογία τη ε, κυρία Κορνέλη εν το θέμα ε, ανθρώπων που μένουν σε άλλη χώρα. Καταλαβαίνω αν μένουν σε άλλο κράτο μέλο, δεν είμαι βέβαια όσον αφορά τι νομικέ πτυχέ. Και τέλος, δεύτερη φορά λέω τέλος, αλλά τέλος πάντων, τροπολογία 50 λέει ε, να παρακολουθεί την... Ε, να ελέγξουν αποτελεσματικά την ενίσχυση που δίδεται σε πολυεθνικέ εταιρείε και για να εγγυηθούν την ε, πραγματοποίηση συνεπού επένδυση για δημιουργία θέσεων εργασία με κοινωνικά δικαιώματα, με σκοπό να αποθαρρυνθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ. Το δεύτερο μέρο νομίζω ότι είναι καλό, το πρώτο μέρο όμω ίσω να να, να, να μην ε, μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν βρίσκω την τροπολογία. Ξέρω ότι η κυρία Κορνέλησεν έχει ε, μία τροπολογία για παράταση της ε, χρονικής περίοδου ε, στους 36 μήνες. Ξέρω ότι η συγγήτρια δεν είναι υπέρ. Κυρία Άρκιν, θα σας σταματήσω διότι μακρηγορείτε. Ε, μπορείτε να έχετε ε, διμερή διαβούλευση με ε, την κυρία Μωρέα. Διότι αλλιώς θα προλάβουμε το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Κορνέλησεν. παρακαλώ να είσαστε τηλεγραφικοί, πολύ σύντομοι. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία ε, εκτός συνεδρίασης. Κυρία Κορνέλησεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Το θέμα με τα προβλήματα για, του Ταμείου ε, ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Νομίζω ότι οι λύσεις που προτείνουμε είναι κάπως διαφορετικές. Όσον αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών ε, και την ε, συντόνιση του χρονικού διαστήματος που θα διατίθεται τα χρήματα, αυτό νομίζω μας βρίσκει σύμφωνος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό βραχυπρόθεσμα, αλλά ίσως μακροπρόθεσμα θα πρέπει να γίνουν πιο θεμελιώδεις ε, αλλαγέ. Αυτό προσπάθησα να το συμπεριλάβω στην τροπολογία μου υπαριθμών 5. Ίσως η κυρία Χάρκιν να έχει δίκιο όσον αφορά την ε, γλωσσική πτυχή. Πολύ ευχαρίστω θα βελτιώσω την τροπολογία αυτή. Πάντως αυτή είναι η γενική μας θέση. Πολλέ τροπολογίε αναφέρονται σε ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού. Προσπάθησα στην τροπολογία 5 να προτείνω να μην επιλέξουμε αμέσως τη λύση αυτή, αλλά να θεσπίσουμε τα κριτήρια να πούμε ότι θέλουμε να είναι πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο και ε, πιο συμπεριληπτικό ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ε, ευφυείς ε, ιδέες και προτάσεις ε, για τις οποίες να μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας όταν αναθεωρήσουν τον κανονισμό όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα της κυρίας Μωρέ, διότι αυτό είναι θέμα που ζήτησαν οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου πρέπει να δημιουργηθεί η ε, η υποδομή για την εφαρμογή εφόσον από τη στιγμή που θα διατεθούν τα χρήματα, διότι τότε ε, μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον μισό έτος μέχρι να ξεκινήσει η παρέμβαση. λοιπόν μιλάμε για κύκλο διετίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει εντός του χρονικού πλαισίου αυτού. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλύτερο να μην, αναφερώ, να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα νούμερα. Πολύ ευχαρίστω θα το αλλάξω αυτό αν, σας, αν ε, βοηθήσει να πετύχουμε υποστήριξη για την τροπολογία αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε κάποιες τροπολογίες για τη συμμετοχή των εργαζομένων ε, στη φάση της εφαρμογής τροπολογίες υπαριθμών 11 και 16. Τον προηγούμενο μήνα 35.000 ευρώ δόθηκαν για τεχνική βοήθεια για να οργανωθεί ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών που ζητούν που κάνουν αίτηση για τη χρηματοδότηση αυτή. Πιστεύω επίση ότι θα πρέπει να του ζητήσουμε να οργανώσουν ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εργαζομένων. Ε, στην Ιρλανδία έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από το μηδέν όσον αφορά την οργάνωση και θα ήταν πολύ κρίμα εάν όλοι θα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Η τροπολογία μου υπαριθμό 48 όσον αφορά τους αλλοδαπούς. Κύριε Κορνέλησεν, θα σας διακόψω. Σας ε, καλώ να κλείσετε την ε, παρέμβασή σας ε, και να τα, ξεκαθαρίσετε τα ζητήματα αυτά διμερώς με την κυρία Μωρέ. Θα μπορούσε η κυρία Μωρέ να προσπαθήσει να Σα υποβάλει προτάσεις, αλλά βρισκόμαστε υπό πολύ πίεση χρόνου. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι το εξή. Έγιναν συζητήσεις στην Επιτροπή προπολογισμού. και Μπορούμε να το σκεφτούμε απόψε, μπορεί να έχουμε προφορική τροπολογία αύριο, αλλά στην Επιτροπή μας υπήρχε συνένεση ότι η έκθεση θα πρέπει να λέει με σαφείς όρους ότι θέλουμε να διατηρήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής. Η απλοποίηση, οι παρεκκλήσεις ε, που θα θεσμιστούν στα πλαίσια της κρίσης ε, θα πρέπει να διατηρηθούν και μετά. Τα δύο αυτά στοιχεία, όταν συζητήθηκε το θέμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, και ξέρω ποια είναι η θέση σας κυρία Ομορά, αλλά... Υπάρχει αυτό στην ε, έκθεση, αλλά στην Επιτροπή Προπολογισμού η συζήτηση θα είναι η ίδια που ήταν κατά τη δημιουργία του Ταμείου. Η δική μας έκθεση θα πρέπει να είναι ε, ακόμα πιο ξεκαθαρή ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό να το έχουμε κατά νου κατά την προσαρμογή του κειμένου. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Κυρία Μωρέ, ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε. Μήπως θα μπορούσα να σας παρακαλέσω να το κάνετε αυτό διμερός, διότι... Ναι, κυρία Πρόεδρε, πράγματι λέει κυρία Μωρέ. Απλά θα ήθελα να καλέσω τι ε, συναδέλφου ε, να σαρθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε όλε τι διαφορετικέ απόψει μα. Euh, ε, ξέρετε, δεν μπορούμε να είμαστε δύο μέρη ταυτόχρονα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε για αυτή την ε, κοινή συνάντηση με την κυρία Τζένσεν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Θα μας παρουσιάσει κυρία Γιάννσεν ε, ε, την έκθεση για το εμπόριο και την απασχόληση στα πλαίσια του διεθνούς εμπόριου. Νομίζω ότι ενδιαφέρει και τις δύο επιτροπές το θέμα. Θα σας δώσω το λόγο και ε, δυστυχώς πρέπει εγώ να αποχωρήσω και θα ε, παραχωρήσω την προεδρία στην κυρία Λίν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στους ε, συντάκτες ε, της έκθεσης. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να συμπροεδεύω εδώ με την ε, κυρία Περές. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα στην Ολομέλεια στο Κοινοβούλιο. Και νομίζω Επειδή αυτό το βιβλίο και αυτή η έρευνα αφορά το εμπόριο και την απασχόληση, είναι πολύ λογικό να συναντιόμαστε εδώ για να ακούσουμε την παρουσίαση του βιβλίου αυτού. I Μπόρεσα να διαβάσω τη σύνοψη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική έρευνα, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, όχι μόνο για την ανάλυση των επιπτώσεων της μείωσης των εμπορικών ροών στην ε, ανεργία και στους μισθούς, αλλά και για τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε για το μέλλον. Για τις απαντήσεις που μπορούν να βρουν οι κυβερνήσεις στο μέλλον, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές κρίσεις Ελπίζοντα με διαφορετικό τρόπο από ότι ο τωρινό. Να συγχαρώ λοιπόν τους συγγραφείς αυτής ε, της ε, τη έρευνα και αυτού του του βιβλίου και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τα συμπεράσματά του τώρα και κυρίως αυτά τα οποία προτείνουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Να δώσω απευθείας λοιπόν το λόγο στην εμπειρογνώμονα από τη Διεθνή Οργάνωση εργασία την κυρία Μαριον Γιάνσεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μορέιρα, την κυρία Λίν για την εισαγωγή και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι εδώ σήμερα. Θα σας παρουσιάσω αυτή τη δημοσίευση, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, τη βλέπετε και στην οθόνη. Είναι ε, έτσι το βιβλίο, έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπό μας. Δυστυχώς ετοιμάσαμε κάποιες διαφάνειες οι οποίες δεν θα φαίνονται στην οθόνη. Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας καθοδηγήσω στην παρουσίαση. Νομίζω ότι έχετε και σχετικά φωτοτυπίε. Ε. Μας ενδιαφέρει το θέμα του εμπορίου και τη ανεργία ε, στην παγκόσμια κρίση, διότι αυτό είναι τμήμα τη συνεχιζόμενης έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις επιπτώσεις τη παγκοσμιοποίηση. Επίσης, ανταποκρίνεται σε, μία, ε, σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό οργανώσεων διεθνών. Ε, το παρουσιάσαμε τη Δευτέρα σε μια σε εναν ολοενα αυξανομενο αριθμο οργανωσεων διεθνων ε το παρουσιασαμε τη δευτερα σε μια διασκεψη με την Παγκόσμια Τράπεζα και είχαμε εκπροσώπου από διάφορε διεθνεί οργανώσει, τον ΟΣΑΤ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση. Το θέμα της παγκοσμιοποίησης λοιπόν και της απασχόλησης ενδιαφέρει όλους ε, αυτή τη χρονική στιγμή, ε, πολλό δε μάλλον λόγω της κλίσης. Προσπαθούμε να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς ε, συνέβη αυτή η κρίση, η οποία ξεκίνησε στον χρηματοοικονομικό τομέα σε μια χώρα, πέρασε στην πραγματική οικονομία, από το χρηματοπιστωτικό τομέα στην πραγματική οικονομία και πώς πέρασε από τη μία χώρα στην άλλη και πώς τελικώς επηρέασε τις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο. Πρόκειται για μια κρίση η οποία εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και δεν ήταν ε, επικεντρωμένη σε μια γεωγραφική περιοχή. Αυτοί οι παράγοντες μετάδοσης λοιπόν ε, ήταν το εμπόριο, γι' αυτό λοιπόν εξετάζουμε το πώς το εμπόριο μετάδοσε την κρίση από τη μία χώρα στην άλλη και πώς επηρέασε την απασχόληση στην κάθε χώρα από εκεί και πέρα. Το εμπόριο ουσιαστικά κατέρευσε κατά τη διάρκεια της κρίσεως. Το εμπόριο ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στην κρίση και ε, μειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ περισσότερο από το ΑΕΠ, ε, ε, έπεσε κατά, περίπου κατά 12% ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ έπεσε κάπου γύρω στο 3% αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία. Και αυτή η τεράστια πτώση οφείλεται στο γεγονός ότι οι χώρες είναι πλέον ε, τόσο ολοκληρωμένες και χρησιμοποιούν παγκόσμιες αλυσίδες προμηθειών. Εάν ένας καταναλωτής σε μια χώρα δεν αγοράσει ένα αυτοκίνητο, αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται η αγορά ε, ελαστικών σε μια χώρα, ε, των μεταλλικών τμήματων σε μια άλλη χώρα και των εξαρτημάτων σε τρίτη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι πλήττονται λοιπόν πολλές χώρες και φυσικά πλήττονται και η απασχόληση λόγω του εμπορίου. Οι επιπτώσεις στο εμπόριο ήταν πολύ σημαντικότερες σε χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο αριθμό εξαγωγών σε τομείς που πλήχτηκαν περισσότερο από την κρίση. Οι τομείς αυτοί ήταν ο τομέας των καυσίμων και των υλικών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, πιο συγκεκριμένα, και επομένως χώρες ε, που ε, δίνουν χάλιβα, για παράδειγμα, στις κατασκευαστικές βιομηχανίες, ε, η Ουκρανία ή η Λιβερία που δίνει ελαστικό για τα ε, ελαστικά των αυτοκινήτων, είχαν σημαντικές πτώσεις στο εμπόριο. Οι κατασκευαστικές εταιρείες και η απασχόληση στο τομέα αυτό μειώθηκε παγκοσμίω. Είχαμε μεγάλη μείωση στι ΗΠΑ, πολύ μεγάλη μείωση και στην Ευρώπη αλλά και στην Ασία. Σε κάποιου άλλου τομεί ε, ε, η απασχόληση ε, άντεξε πολύ περισσότερο στην Ασία, αλλά σημειώσε πολύ μεγάλη πτώση στι ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Δηλαδή κυρίω στο κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των οικοδομών και στον τομέα του εμπορίου εν γέννη. Το εμπόριο θεωρούμε ότι πλήχθηκε. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση εκδηλώθηκαν με λιγότερες θέσεις εργασίας αλλά και με χαμηλότερους μισθούς, χαμηλότερο ε, αριθμό ωρών εργασίας και ακριβώς επειδή υπήρχαν επιπτώσεις στην απασχόληση ε, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε και να μετρήσουμε τι συνέβη στις αγορές και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Σε μια χώρα ε, πλήττονται οι θέσει εργασία, σε μια άλλη χώρα πλήττονται οι μισθοί και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι τελείω διαφορετικά και υπάρχουν γενικευμένα μηνύματα τα οποία δεν μπορούμε όμω να αποστείλουμε γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώ κάνει το εμπόριο στην απασχόληση. Για να το κατανοήσουμε αυτό πιο καλά και πιο διεξοδικά, τι ρόλο έπαιξε το εμπόριο στην απασχόληση, εξετάσαμε κάποιες χώρες πιο αναλυτικά κυρίως σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες και σε μεγάλο βαθμό κατόπιν ετήσεως των χωρών αυτών που ζήτησαν από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας να του δώσουν κάποιες συμβουλές για την μετρίαση της κρίσης και να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τι συνέβη με την απασχόληση ε, στις χώρες τους. Είχαμε την Ουκρανία, τη Λιβερία, την Ουγκάντα, την Ινδία, την Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και την Αίγυπτο. Εκεί έγινε η αξιολόγηση του τι ακριβώ συνέβη ε, με την απασχόληση λόγω του εμπορίου. Και θα σας δώσω και κάποια στοιχεία από τις χώρες αυτές. Μπορεί να νομίζετε ότι οι χώρες αυτές πόρα απέχουν από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι μεν, αλλά κάποια από τα στοιχεία τα οποία διαπιστώσαμε έχουν σημασία και για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στην Ουκρανία μας ζητήθηκε να εξετάσουμε το ρόλο που έπαιξε η συγκέντρωση των εξαγωγών. Η Ουκρανία έζησε ένα οικονομικό σοκ, αλλά πλήχθηκε και από τις ε, μειώσεις ε, στις μεταλλουργικές εξαγωγές. Μα ζητήθηκε λοιπόν να του βοηθήσουμε να εξηγήσουν τι συνέβη και να του δώσουμε και κάποιε ε, συμβουλέ για να βελτιώσουν την ε, διαφοροποίηση στι εξαγωγέ. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η Ουκρανία πριν από την κρίση ε, εξήγαγε προϊόντα στους περισσότερο πληθέντες τομείς αλλά και στις περισσότερο πληγήσεις περιοχές. Κυρίως εξάγει στις χώρες της κοινοπολιτείας και στη Δυτική Ευρώπη. Και οι δύο περιοχές πλήχθηκαν πολύ σοβαρά από την κρίση, έπεσε το ΑΕΠ, μειώθηκε η ζήτηση, μειώθηκαν οι εισαγωγές. Η Ουκρανία εξάγει πολύ λίγα στην Ασία, κυρίως στην Κίνα και στην Ινδία και ε, πολύ λίγα σε χώρες όπως την Βραζιλία. Το γεγονός λοιπόν ότι ήταν ε, συγκεντρωτική προσέγγιση του ήταν όχι μόνο στα προϊόντα αλλά και ω προ μια προσπάθεια στη διαφοροποίηση των εξαγωγών και προς άλλες γεωγραφικές περιοχές. Επίσης ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οργανισμοί ε, που θα βοηθήσουν στις χώρες να κάνουν, τη χώρα να κάνει ταυτόχρονα επενδύσεις σε κεφάλαια αλλά και σε δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν τη χώρα να αναβαθμίσει το επίπεδο των εξαγωγών της και να περάσει και σε άλλους τομείς για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί περισσότερο η Ουκρανία, ακριβώς επειδή ήταν πολύ μεγάλο το πλήγμα, έχασε ε, πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Υπήρχαν κάποιους ε, τομείς στους οποίους οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 15 ή 16%. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Ένας από τους τομείς στον οποίο χάθηκαν πολλές ε, ε θέσεις εργασίας ήταν στα ορυκτά προϊόντα ε, που είναι μη μεταλλικά. Εδώ δεν έχουμε πολλές εξαγωγές, αλλά χάθηκαν πάρα πολλές θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό. Ο τομέας αυτός όμως δίνει ε, εισαγωγικά προϊόντα στον τομέα, τομέα που εξάγει, δηλαδή εισάγει προϊόντα για τον τομέα της μεταλλουργίας. Επειδή μειώθηκαν οι εξαγωγές, ε, δεν χρειάζονταν πλέον εισαγωγές προϊόντων, επομένως μειώθηκαν και οι θέσεις εργασίας. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι η οικονομία πλήχθηκε στον τομέα της μεταλλουργίας, ε, είχαμε κάποιες επιπτώσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε μη εξαγωγικού τομές. Είχαμε έμεσες λοιπόν επιπτώσεις που ήταν πάρα πολύ σοβαρές και αυτό αποτελούσε ένδειξη του γεγονότος ότι πρέπει να εξετάσουμε και τις έμεσες επιπτώσεις. Διότι αυτό που γίνεται κατά τη διάρκεια μιας εμπορικής κρίσης είναι ότι συνήθως οι κυβερνήσει θέλουν να βοηθήσουν τον τομέα που πλήττεται, δηλαδή τον εξαγωγικό τομέα. Αλλά αν δώσουμε για παράδειγμα επιδοτήσει στην ενέργεια για τι εξαγωγέ, αλλά ο τομέα δεν μπορεί να εξάγει περισσότερο γιατί κανένα δεν αγοράζει τα προϊόντα του, οι προμηθευτέ εξακολουθούν να πλήττονται και εξακολουθούν να χάνονται θέσει εργασία. Το να κατανοήσουμε λοιπόν τι έμεσε επιπτώσει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο κάναμε στη, στη Νότια Αφρική και δεν θα μιλήσω για την Αίγυπτο, θα πάω στον πίνακα για την Νότια Αφρική. Στη Νότια Αφρική κάναμε πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα, χρησιμοποίησαμε μεγάλα, ε, μεγάλες ομάδες δεδομένων και είχαμε και ποσοτικά μοντέλα γιατί έχουμε τέτοια μοντέλα για χώρες όπως η Νότια Αφρική. Ε, είναι λίγο υπερβολικά από θεωρητική σκοπιά σε αυτά τα μοντέλα, αλλά μας επιτρέπουν να μετρήσουμε πολύ, με πολύ μεγαλύτερη ε, ακρίβεια ε, ποια είναι η επίπτωση σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, στο εμπόριο επί και μας επιτρέπει να μετρήσουμε και να κατανοήσουμε πώς το πρόβλημα μετακινείται από τον εξαγωγικό τομέα στους άλλους τομείς. Ένα από τα πιο σημαντικά μας ευρήματα είναι ότι αυτό το οποίο μετρήσαμε με αυτό το μοντέλο και αυτό το οποίο εκτιμήσαμε ήταν απώλεια περίπου 900.000 θέσεων εργασίας στην Νότια Αφρική, που είναι περίπου αυτό που παρατηρήσαμε, αλλά 390.000 από αυτές τις 900.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν είναι από τις έμεσες επιπτώσεις και κυρίως από την επίπτωση στο εισόδημα. Τι σημαίνει η επίπτωση στο εισόδημα. Σημαίνει ότι λόγω εξαγωγών χάνονται θέσεις εργασίας, έχουμε χαμηλότερους μισθούς και επομένως αγοράζουν λιγότερα λούχα, ε, ξοδεύουν λιγότερα, πηγαίνουν σε λιγότερα εστιατόρια και αυτό φυσικά πλήττει και άλλους τομείς, διότι αυτές οι απώλειες πλήττουν και άλλου τομεί στην οικονομία και διαπιστώνουμε ότι αυτές οι έμεσες επιπτώσεις είναι τεράστιες είναι περίπου το μισό των συνολικών επιπτώσεων, δηλαδή το 50% είναι έμεσες επιπτώσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χάραξη της πολιτικής, διότι αυτά τα οποία γίνονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων είναι για να αντιμετωπίσουμε και τις έμεσες επιπτώσεις. Επίσης, ε, διαπιστώσαμε ότι έχουμε πολύ καλή προσέγγιση των στοιχείων αυτών με τα μοντέλα και διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά υλοποιούνται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν, δεν χρειάζεται ένας χρόνος, μέσα σε λίγους μήνες γίνονται. Παρά το γεγονός ότι το σοκ είναι προσωρινό, ακόμα και αν είναι μια κρίση που διαρκεί ένα χρόνο και ακόμα και αν πλήττει μόνο ένα τομέα, κατά πάσα πιθανότητα θα εξοπλωθεί σε όλη την οικονομία πολύ γρήγορα και αυτή η εξάπλωση είναι αυτή που προσπαθούμε να αποφύγουμε με τα μοντέλα μπορέσαμε να εξετάσουμε και ποιοι είναι αυτοί που πλήττονται σε μια οικονομία από το σοκ. Ποιο χάνει θέση εργασία, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, αυτοί με υψηλέ δεξιότητε, αυτέ με λίγε δεξιότητε, οι άνδρε, οι γυναίκε. Ε, με το μοντέλο της Νοτιοαφρικής το ε, εξετάσαμε αυτό και το ίδιο κάναμε και με τη μελέτη για τη Βραζιλία. Στην Νότια Αφρική διαπιστώσαμε ότι είναι κυρίως ε, αστικά νοικοκυριά αυτά τα οποία πλήττονται. Είναι περισσότερα από τα ε, ε, νοικοκυριά της Υπέθρου. Και διαπιστώσαμε επίσης ότι μεταξύ των αστικών νοικοκυριών και των νοικοκυριών της Υπέθρου είχαμε απώλειες σε όλες τις κλίμακες. Και στους πλούσιους και στους φτωχούς και στου λιγότερο πλούσιους και στου λιγότερου φτωχούς. Οι πλούσιοι είναι αυτοί που πλήχθηκαν περισσότερο ε, αυτοί που είναι καλύτερα δηλαδή ενσωματωμένοι στην άμεση οικονομία ε, χτυπιούνται πιο πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, λόγω των μοντέλων μπορέσαμε να δούμε και πώς ε, ε κινήθηκαν αυτοί που ε, έχουν μισθούς, ε, αυτοί που έχουν κεφάλαια και διαπιστώσαμε ότι όσοι ε, κερδίζουν ε, ψηλά κεφάλαια χτυπήθηκαν πολύ πιο άμεσα, αλλά επίσης είχαμε και πολύ μεγάλο πλήγμα για αυτούς που έχουν χαμηλούς μισθούς. Επομένως είχαμε τα δύο άκρα, τους πολύ πλούσιους και τους πολύ φτωχούς. Ενδιάμεσα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο άσχημα, ε, κυρίως για τους μισθωτούς. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξαγωγική δομή που έχουμε σε χώρες όπως η Βραζιλία για παράδειγμα, όπου περιμένουμε να έχουμε μια βιομηχανία που βασίζεται σε ε, προϊόντα εντατική ε, παραγωγής. Σε άλλες χώρες όπως στην ε, Ουκρανία οι μεσαίου εισοδήματος μισθωτοί πλήχθηκαν. Με τη μελέτη της Βραζιλίας μπορέσαμε να εξετάσουμε και το προϋπολογισμό της κυβέρνησης πώς ο προϋπολογισμός της, ε, της κυβέρνησης Βραζιλίας ε, επηρεάστηκε από την κρίση. Κάναμε μία προσωμείωση και μετρήσαμε ποιες ήταν οι αναμονόμενες απώλειες ε, στους δασμούς εισαγωγών για τη Βραζιλία κατά τη διάρκεια της κρίσεως, ποια θα ήταν η απώλεια στα εισοδήματα από τη φορολογία λόγω της πτώσης του ΑΕΠ και τα εισοδήματα από τη φορολογία. Και είπαμε έστω ότι η Βραζιλία θέλει να κάνει έναν ισορροπημένο προπολογισμό και θέλει να αυξήσει τους άμεσους ε, φόρους ε, εισοδήματος για να ε, εξισορροπήσει τα πράγματα από τις απώλειες που είχε. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η Βραζιλία θα έπρεπε να αυξήσει τους άμεσους φόρους εισοδήματος κατά 5% για να εξισορροπήσει την απώλεια εισοδήματος. Και γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Είναι γιατί η Βραζιλία είναι μεγάλη χώρα, ε, δεν έζησε ένα οικονομικό σοκ, αλλά ε, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το λάβουμε υπόψη στο μοντέλο μας. Δεν μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη επίσης και την, ε, ε, τα πακέτα για κίνητρα και εξετάσαμε μόνο την απώλεια εισοδήματο λόγω της επιβράδυνσης. Και για να γίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αυξηθεί ο φόρος εισοδήματο κατά 5%. Νομίζω ότι αυτό αναπαριστά πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη είναι η πίεση στον κυβερνητικό προπολογισμό λόγω του σοκ που υπέστημεν όλοι προσφάτως. Στη Λιβερία, μια χώρα πολύ διαφορετική από τις ευρωπαϊκές χώρες, ε, δεν μπορούσαμε να έχουμε μοντέλα, δεν είχαμε κανένα στοιχείο και για να ε, εξετάσουμε τις επιπτώσεις στην απασχόληση σε μια τέτοια χώρα είναι να πάμε στη χώρα να βρείτε εθνικά δεδομένα, οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε για, για να έχετε μια αίσθηση του τι συνέβη με την απασχόληση πρέπει να μιλήσετε με τους ενδιαφερομένους και με τους κοινωνικούς εταίρους και αυτό έκανα γιατί μιλάω για τη Λιβερία παρά το γεγονός ότι διαφέρει τόσο πολύ με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι στη Λιβερία είχαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η τα που διαπιστώσαμε ε, στις ε, κρίσεις ε, και λόγω της διακύμασης των τιμών των τροφίμων πριν από την κρίση πώς μπορούν να επηρεάσουν μια χώρα και την ανάπτυξή της μακροπρόθεσμα επειδή ακριβώς υπήρχαν μεγάλες διακοιμάνσεις, οι επιχειρήσεις περίμεναν προκειμένου να κάνουν επενδύσεις. Αυτό γιατί ε, περίμεναν να δουν τι θα γίνει και έτσι είχαμε με λιγότερη ανάπτυξη, που σημαίνει ότι στη Λιβερία ε, υπήρχαν προβλήματα. Αυτοί που δεν είχαν εισοδήματα σκεφτόντουσαν να μεταναστεύσουν και έφτασαν και τα παιδιά του από το σχολείο, κυρίω τα κορίτσια. Είχαμε μικρότερε προσδοκίε για το μέλλον, μικρότερη ανάπτυξη. Επίση, μπορεί να απληχθεί και η ίδια κυβέρνηση. Στη Λιβερία, η κυβέρνηση διαπραγματευόταν ε, κάποιε συμφωνίε με ε, ξένε πηγέ. Είχαμε εκχωρήσεις για τα ορυχεία, και επειδή ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα και χρειαζόντουσαν κατεπηγόντω τη ε, κατέληξαν σε πολύ άσχημε συμφωνίε για τη Λιβερία και επομένω υπήρχαν πρόβληματα και λιγότερα εισοδήματα για τη χώρα στο μέλλον. Πρόκειται για κάτι το οποίο γνωρίζουν οι χώρε εδώ και αρκετό καιρό. Τα, οι διακυμάνσει, η ευμεταβλητότητα είναι πολύ σοβαρή και για να μειώσουμε τα ποσοστά που έχουμε ε, δει στη πρόσφατη οικονομία, ε, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Εξετάσαμε διάφορους τρόπους να εξετάσουμε, να δούμε τις επιπτώσεις του εμπορίου. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, κυρίως ε, στα πλαίσια ε, ενός μεγάλου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέγεται Unsessing and Addressing the Employment Effects of Trade και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δούμε τι επιπτώσεις έχουμε στην απασχόληση από το εμπόριο σε χώρες που θεωρούμε στόχο. Εργαζόμαστε στο συγκεκριμένο τομέα με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τα θέματα της πολιτικής τώρα, τι κάναμε. Στη διάρκεια της κρίσεως και ακόμα και πριν από την κρίση ε, ε, μας είχε ζητηθεί να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στη χάραξη πολιτικής. Επομένως, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα θέματα της εργασίας, ε, του εμπορίου, είναι συνεκτικές και δεν είναι αντικρουόμενες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο είναι να δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να έχουμε συνεκτικά μηνύματα στη διάρκεια της κρίσεως, ε, όπως η κρίση που αντιμετωπίσαμε, και από πλευράς εμπορίου αλλά και από πλευράς απασχόλησης. Επομένως, αναλύσαμε κάποιες συμβουλές ε, πολιτικής που δόθηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε, για παράδειγμα, τις ε, παγκόσμιες θέσεις εργασίας και τις συμβουλές που δίνονται και κάποιες συστάσεις από άλλους οργανισμούς, ε, κυρίως τον ΠΟΕ. Και είδαμε κατά πόσον αυτά τα μηνύματα πολιτικής συνάδουν ή είναι αντικρουόμενα. Και από τις δύο πλευρές υπήρχε συμφωνία και υπάρχει γενικά συμφωνία ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης σε διεθνές επίπεδο ότι δεν θα πρέπει να ε, πέσουμε στην παγίδα του φαύλου κύκλου του προστατευτισμού. Αυτό δεν θα βοηθήσει ούτε την παγκόσμια οικονομία ούτε το εμπόριο. Και υπάρχουν προειδοποίησεις κατά του προστατευτισμού και αυτά προέρχονται και από άλλους διεθνούς οργανισμούς, κυρίως από τον ΠΟΕ. Στη διάρκεια της κρίσης και στην αρχή της κρίσης ε, υπήρχαν πολλοί φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση θα επηρεάσει το εμπόριο, διότι οι εξαγωγείς δεν θα είχαν πρόσβαση σε ε, πιστώσει εξαγωγών και αυτές είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσει να πληρώσει κάποιους εξαγωγέ. Επομένω, υπήρχε έκκληση για βοήθεια από τις κυβερνήσεις για τις ε, πιστώσει εξαγωγών και οι χώρε του G20 ε, δέσμευσαν ένα ποσό 250 δι για τη χρηματοδότηση του εμπορίου. Διαπιστώσαμε και στην Ουκρανία αλλά και στο Μαρόκο ότι ε, ναι, μεν οι χώρε ε, διέθεταν κονδύλια για το εμπόριο, αλλά οι επιχειρήσει δεν το χρησιμοποιούσαν. Και γιατί αυτό, γιατί κανεί δεν ήθελε τα προϊόντα του. Επομένω δεν μπορούσαν να εξαγάγουν προϊόντα. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την εξαγωγή, αλλά ότι δεν ήθελε κανεί τα προϊόντα του. Δεν υπήρχε ζήτηση και επομένω ε, δεν ε, τίθεται το θέμα χρηματοδότηση. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο συμπέρασμα για πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Επίσης εξετάσαμε ε, την κρίση σε τομεακές πολιτικές. Και γιατί εξετάσαμε τις πολε... τομεακές πολιτικές. Οι τομεακές πολιτικές ε, στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς ή σε συγκεκριμένους επιχειρήσεις. Επί παραδείγματι, ο μεταλλουργικός τομέας στην Ουκρανία ή κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς που πλήχθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτές οι πολιτικές δεν είναι πολύ ευπρόσδεκτες τις συμφωνίες του ΠΟΕ. Υπάρχει μια συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα ε, μέτρα αντιστάθμισης, όπου οι επιδοτήσεις απαγορεύονται και οι επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους τομείς θεωρούνται ε, ότι ε, μπορεί κάποιο να τι αντικρούσει. Μπορεί δηλαδή ένα κράτο μέλο να πει ότι σταματήστε, δεν μα αρέσουν αυτέ οι πολιτικέ. Οι πολιτικέ εμπορίου θεωρούνται ότι στευρώνουν το εμπόριο και δημιουργούν προβλήματα, είναι αναπιθύμητε. Και αυτό προκύπτει και από τα μηνύματα του G20 στην έκθεση η οποία απεστάλλει ε, στο G20. Βάσει του Συμφώνου των Παγκοσμίων Θέσεων Εργασίας ε, υπάρχει κάποια υποστήριξη. Εδώ έχουμε κάτι αντικρουόμενο. Ναι, μεν ε, ε, υποστηρίζεται από τη μία πλευρά, το εμπόριο δεν τα υποστηρίζει. Η ε, στο G20 είπε ότι για λόγους διακρίσεων θα πρέπει να κάνουμε ένα καταμερισμό μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν τις πολιτικές του εμπορίου και αυτές που υποστηρίζουν το ΑΕΠ. Θα πρέπει να υπάρχουν δηλαδή αποσύνδεση ε, στις πολιτικές που υποστηρίζουν το κεφάλαιο και θα πρέπει να αλλάξει σε σχέση με αυτά που ε, υποστηρίζουν την εργασία. Υπήρχε μια συζήτηση του ΩΣΑ που εξηγούσε γιατί μέτρα που στοχεύουν στην απασχόληση κατά τη γνώμη τους είναι πιο χρήσιμα σε κατάσταση κρίσης ε, από ότι τα μέτρα που στοχεύουν αλλού, για παράδειγμα, την πλευρά του κεφαλαίου διαφόρων τομέων. Μία εξαίρεση σε αυτήν την τομεακή συζήτηση είναι η υποδομή. Η υποδομή ε, ήταν το επίκεντρο προσοχής σε πολλές χώρες. Πολλά χρήματα έχουν δαπανηθεί σε μέτρα υποδομής. Ε, και στα πλαίσια του ΠΟΕ ε, δεν θεωρούμε τα μέτρα αυτά ότι στρεβλώνουν το εμπόριο. Η καλύτερη υποδομή έχει την ε, δυνατότητα να μειώσει το κόστος ε, των μεταφορών ε, και έτσι να διευκολύνει το εμπόριο. Είναι λοιπόν καλές για το... είναι καλά τα μέτρα αυτά για το εμπόριο. Ε, τέλος, εξετάσαμε και άλλα μέτρα, διατομεακά μέτρα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα. Μέτρα δηλαδή που δεν στοχεύουν σε συγκεκριμένο τομέα ή σε συγκεκριμένη επιχείρηση αλλά που στοχεύουν σε συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τους ανέργους, τους στοχούς, τους νέους ή τους ηλικιωμένους. Δεν έχουν λοιπόν σαν στόχο ε, κάποιον παραγωγικό τομέα, ε, αλλά στοχεύουν σε συγκεκριμένε ε, ομάδε του πληθυσμού. Αυτά τα μέτρα δεν θεωρείται ότι στρεβλώνουν το εμπόριο και μπορούν να έχουν και και μπορούν να αντιμετωπίσουν και, τα άμεσα και, τα, και τις άμεσες και τις άμεσες ε, συνέπειες ε, κάποιου κλονισμού στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας άνεργος ε, λαμβάνει επίδομα επειδή είναι άνεργος, άσχετα από άλλους παράγοντες. Η δουλειά του ΔΟΕ αλλά και της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνει ότι οι διατομιακές πολιτικές όπως αυτές ε, είναι πολύ αποτελεσματικές σε περίπτωση εξωτερικών κλονισμών, ιδιαίτερα αν υπάρχουν πριν την κρίση. Για παράδειγμα, υπήρχε ένα πρόβλημα στη Βραζιλία, το οποίο παρήχε εισοδήματα σε φτωχέ ε, οικογένειε. Κατά τη διάρκεια τη χρήση, περισσότεροι άνθρωποι έπεσαν στην ε, ένδια ε, και λάμβαναν έτσι ε, χρήματα. Ε, η κυβέρνηση μπόρεσε να αλλάξει τη φύση του προγράμματος, να βελτιώσει την πρόσβαση για τις οικογένειες. Σε τη στιγμή που ήδη υπάρχει ένα μέτρο μπορεί κανείς εύκολα να το τροποποιήσει. Το να το οικοδομήσει κατά τη διάρκεια μιας κρίσης είναι πολύ δύσκολο, διότι αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. Οι διατομιακές πολιτικές λοιπόν συχνά είναι πολιτικές ε, του τύπου κοινωνικής, συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Είναι λοιπόν πολύ αποτελεσματικά κατά διάρκεια κρίσεων. Αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια τη παρούσα κρίση, ε, αλλά ε, και σε άλλες κρίσεις όπως για παράδειγμα η Ασιατική, που υπήρχε πριν κάποια χρόνια όσον αφορά του ε, κλονισμού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης ήταν πολύ ε, σημαντικέ ε, σε όλες τις χώρες που εξετάσαμε. Σε κάποιες χώρες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Είδαμε ότι οι έμεσε συνέπειε στην απασχόληση είναι πολύ σημαντικέ και ότι φαίνονται πολύ γρήγορα. Το να επικεντρωθούμε λοιπόν μόνο στην πλευρά του εμπορίου δεν θα καλύψει το σύνολο του προβλήματος. Επίσης διαπιστώσαμε ότι ε, επηρεάζεται η κατανομή, το πώς όμως γίνεται αυτό εξαρτάται από την χώρα και από το τι εξάγει η χώρα. Η αστάθεια και οι κλονισμοί των τελευταίων ετών μπορούν να έχουν ε, μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξη ε, λόγω των συνεπειών στην, στις επενδύσεις. Σε επίπεδο πολιτικής ε, πιστεύω ότι αυτό που κάναμε είναι χρήσιμο εάν θέλει κανείς ε, να βελτιώσει την συνοχή των ε, μέτρων πολιτικής σε διάφορους τομείς. Έχει επικροτηθεί η προσπάθειά μας από συναδέρφους σε, άλλες, σε άλλους διεθνούς φορείς. Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι τα άτομα που θέλουν προστασία ε, από τις ε, κρίσεις που είδαμε τα τελευταία χρόνια και που ε, συχνά σε ατομικό επίπεδο έχουν σοβαρές συνέπειες. Είδαμε ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας όπως συστήματα επιδόματος ανεργίας ή άλλων κοινωνικών εισοδημάτων είναι, που στοχεύουν σε συγκεκριμένε πληθυσμιακέ ομάδε, για παράδειγμα, είναι πολύ αποτελεσματικά και δεν στερβελώνουν το εμπόριο. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μας, αποτελούν μια πολιτική φιλική ως προς ε, την συνοχή. Τα μέτρα αυτά στοιχίζουν χρήματα. Τα περισσότερα μέτρα που λαμβάνονται κατά διάρκεια μιας κρίσης ε, απαιτούν ε, πόρους. Γι' αυτό το να οικοδομηθούν ε, στέρεοι κρατικοί προπολογισμοί κατά τη διάρκεια ε, καιρών ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε ε, πώς επηρεάζεται αρνητικά ο κρατικός προπολογισμό σε εποχέ κρίσης. Εμείς θα προτείναμε η ανάγκη για δημιουργία ισχυρών προϋπολογισμών να μην, αποτελέσουν, να, να μην οδηγήσουν σε, σε ε, θυσία των ε, κοινωνικών ε, συστημάτων, των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, διότι όταν χτυπήσει η επόμενη κρίση θα είναι πολύ αποτελεσματικά μέτρα κατά τη διάρκεια της επόμενης κρίσης και φιλικά, σχετικά με την παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Θα απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσίαση αυτή για όλους μας. Λυπάμαι πολύ που είναι τόσο περασμένη η ώρα δεν ε, έχουμε πολλούς βουλευτές εδώ, αλλά σίγουρα θα φροντίσουμε όλοι οι βουλευτές να λάβουν αντίγραφο της παρουσίασής σας, που θα είναι πολύ χρήσιμη. Έχω έναν-δύο μιλητές ε, προτού να... Ε, ε προτού να να δώσω το λόγο στον κύριο Κοφεράτη. Θα ήθελα να συγχαρώ το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για την εξαιρετική δουλειά του που μας δίνει επιχειρήματα αλλά και στοιχεία, δεδομένα, ε, στοιχεία αξιολόγησης πολύ συγκεκριμένα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για να διασκεδάσουν κάποιους μύθους που αρχίζουν να κυκλοφορούν. Από τη μελέτη βλέπουμε ότι αντιθέτως με αυτό που υποστηρίζουν οι πολλοί, η κρίση χτύπησε πολύ βαριά όλες τις χώρες του κόσμου. Είμαστε συνηθισμένοι λίγο, διότι είναι λίγο ε, παρανοϊκός ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Θεωρούμε ότι η, χρήση, η κρίση που γεννήθηκε στον πιο καπιταλιστικό ε, λαό της Ευρώπης, στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, ε, εξαπλώνεται στις χώρες που έχουν κάποιες ομοιότητες με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Δεν είναι αλήθεια όμως και οι πιο ευάλωτες χώρες ε, πλήχθηκαν ε, πάρα πολύ. Και αυτό φυσικά ε, καταστρέφει ένα σενάριο στο οποίο υπάρχουν στοιχεία ε, παγκόσμιας φτώχειας. Όλοι βρίσκονται σε δυνότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν. Έχει χαθεί πλούτο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ε, από αυτά που μας παρουσιάσατε πάρα πολύ καλά, εντάθηκαν και κάποιες διαφορές και κυρίως κάποιες ανισότητες, οι οποίες αναπόφευκτα θα έχουν συνέπειες και στην επιθυμητή φάση της ανάκαμψης, που μεταξύ άλλων δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει και τι διαστάσεων θα είναι και θα χρειάζεται και μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να μην εντιαθούν αυτές οι διαφορές οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της κρίσης, ίσα ίσα ε, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τους δύο ε, πόλους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι αναφερθήκαμε και στην οικονομική πολιτική και όχι μόνο στην πολιτική εγκαίνη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνει είναι να μην υποχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση του προστατευτισμού ως ε, λύση της χρήσιμης υπεράσπισης των ατόμων. Χρειαζόμαστε μία ρύθμιση μεν στην αγορά, αλλά χρειαζόμαστε αγορά. Εντός αυτής της αγοράς η εργασία θα πρέπει ε, να ξαναλάβει την αξία που έπρεπε να έχει από ιστορική σκοπιά, κυρίως την κοινωνική της αξία. Και για να έχει κοινωνική αξία η εργασία θα πρέπει να, οδηγεί, να συγγνώμη, ένα εισόδημα το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Κατόπιν υπάρχει σημασία της κοινωνικής προστασίας. Τώρα τελευταία αναφερθήκατε στο θέμα της πρόνοιας. Αλλά είναι προφανές ότι τα άτομα τα οποία δεν τα υπερασπίζεται κάποιος στην κοινότητά του είναι τα πιο ευέλωτα και είναι και τα πιο... Ε, προβληματικά, διότι εκεί που δεν υπάρχει προστασία, η αγορά εργασίας είναι ο μόνος χώρος στον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν μία αλλαγή ώστε να πάρουν αυτά που δεν τους διασφαλίζει το κράτος. Ε, την ε, ε, περίθαλψη όταν αρρωσταίνουν, την παιδεία για τα παιδιά τους, το να ζήσουν μια αξιοπρεπή τρίτη ηλικία, όλα αυτά είναι κοινωνική πρόεμνια. Εμένα με φοβίζει κάτι, γι' αυτό ακριβώς με ενδιαφέρει και πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας. Έτσι όπως έχει κατάσταση και δεδομένων και των δυναμικών που θα ακολουθήσουν. Φοβάμαι ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει μια δραστηριότητα μεγάλων εμπορικών ανταλλαγών και στον τομέα των υπηρεσιών, στους οποίους το κυρίαρχο ε, μοντέλο θα βασίζεται στο κόστος, αλλά επίσης για τη μείωση του κόστους ε, αμφισβητούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, παιδιών. Η παιδική εργασία, το να μην μπορεί κάποιος να έχει συλλογική εξπροσώπηση και να οργανώνεται και να μην θεωρούνται θεμελιώδη δικαιώματα, κάποια δικαιώματα που αφορούν στους εργαζομένους. Μήπως λοιπόν τώρα θα έπρεπε ως επιχείρημα συζήτησης να ξαναθέσουμε το θέμα της κοινωνικής ρήτρα. Όχι όμως όπως προτάθηκε πριν από κάποιες δεκαετίες, αλλά με την ε, σύνδεση της αμεβαιότητας. Οι χώρες ε, που είναι πιο φτωχές ε, ζήσαν πάντα την κοινωνική ρήτρα ως ε, μια προσπάθεια να τους εκμεταλλευτούν οι πλουσιότερες χώρες και να τους ε, επιβάλλουν όρους και να τους υποχρεώνουν να εξάγουν προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Ίσως, εάν έχουμε τη ρήτρα αυτή με αυτή την υποχρέωση της αμοιβαιότητας και αυτό το καινοτόμο στοιχείο, να μπορέσουμε να έχουμε ε, κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ για να προλάβουμε τις απαντήσεις. Παρακαλώ ε, να είστε σύντομοι με τις ερωτήσεις. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Ε, το θέμα της κοινωνικής προστασίας ε, και τη χρήση αυτής της έννοιας ως βασική γραμμή είναι κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανοίγει ευρύτερε προοπτικές. Θα υπάρξει όμως παρακολούθηση για να δούμε ποιες θα είναι οι ενδυνάμει επιπτώσεις ελπίζουμε ότι θα νορθωθεί η οικονομία ε, ναι, ε, και θα δούμε ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν στους διάφορους τομείς. Ε, και βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες έχουν πληγεί περισσότερο οι φτωχότεροι. Άρα πώς θα τους στηρίξουμε κυρίως στα πλαίσια των στόχων της χιλιετίας. Η Λιβερία, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και πιστεύετε ότι αυτό έχει επιπτώσεις ε, στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τις ε, φτωχότερες ε, χώρες σε αυτή την περίοδο κρίσης. Και πάλι εδώ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η Λιβερία σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Δηλαδή επειδή χρειάζεται τώρα χρήματα κλείνεται μια συμφωνία που δεν είναι όμως ευνοϊκή και έτσι ε, υπονομεύεται τις ε, μελλοντικέ προοπτικές σας χώρα. Έχω και άλλες ερωτήσεις αλλά θα περιοριστώ σε αυτές. Ο κύριος Σέρκας. Πολύ σύντομα, καταρχάς να σας εγχαρώ για τη δουλειά σας και να σας ενημερώσω ότι θα γίνει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ο Ρίτσαρντ Φάμπερ, ε, ο σοσιαλιστής ευρωβουλευτής που είναι αρμόδιος για αυτή την έκθεση, δεν είναι εδώ, αλλά θα τον ενδιαφέρει σίγουρα να δει το σύνολο της έκθεσης. Θα κάνουμε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την εξωτερική διάσταση και να δούμε πώς μπορούμε να υποστηριχθούμε ε, ώστε το κοινωνικό μοντέλο να παγιωθεί στις διεθνείς οργανώσεις και να συνεχιστεί για ε, να διαπιστώσουμε ότι αυτό που είναι καλό για μας είναι καλό για όλους, διότι όλοι ε, στο ίδιο καράβι πλέουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να έχουμε όλοι σας την έκθεση. Αναφερθήκατε στην ιστοσελίδα και θα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τα στοιχεία αυτά για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Μάλιστα και ο κύριος Μορέιρα. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συντάκτες της έκθεσης. Τρεις παρατηρήσεις. Ε, υπάρχει ευρύτατα ε, η αντίληψη σχετικά με το πόσο αρνητικά επηρεάζει την απασχόληση, η οικονομική κρίση. Συχνά ακούμε εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και αλλού πως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες παρότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ε, κρίση, ε, πλήττονται σφοδρότερα από όλες οι υπόλοιπες. Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις όμως για το αντίθετο, ότι επλήγησαν οι πλουσιότερες χώρες στον τομέα της απασχόλησης να κάνουμε μια σύγκριση με την Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη, καταλήγουμε σαφέστατα σε αυτό το συμπέρασμα. Δεύτερον, αποδεικνύει η έκθεση ότι η καλύτερη απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης ε, στην απασχόληση και τη μείωση της απασχόλησης και τη μείωση των μισθών. Φυσικά δεν είναι ο προστατευτισμός. Ούτε και η τεχνητή διοικητική δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μόνο τα μέτρα κοινωνικής προστασίας που θα δώσουν έπλογο εισόδημα στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι μια σωστή απάντηση. Τρίτον, το άνοιγμα στο εμπόριο τι σημαίνει έκθεση στην, ε, στον ανταγωνισμό και στην κρίση. Φυσικά ε, η κρίση στις εμπορικές συναλλαγές δεν συμβαίνει σε αυτάρκης οικονομίες. Πιστεύω πραγματικά πως ε, μας δείχνει η ιστορία ότι δεν υπάρχει δημιουργία θέσεων απασχόλησης αν δεν υπάρχει άνοιγμα στο εμπόριο. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια χώρα που να κατάφερε να έχει μια ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης χωρίς να ανοίξει την αγορά της. Ε, το εμπόριο και η ανάπτυξη δεν είναι αντικρουόμενε έννοιε. Το αντίθετο, χωρί εμπόριο δεν υπάρχει ανάπτυξη. Μπορεί να υπάρξει εμπόριο χωρί ανάπτυξη, αλλά αν ε, συνδυάσουμε τα δύο, θα γίνει σημαντικός μοχλός το εμπόριο για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μεγαλύτερη ευημερία. Ευχαριστούμε, λέει η κυρία Λίνε. Θα δώσω το λόγο για λίγο στην κυρία Γιάνσεν για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, λυπάμαι, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πολλοί θα προτιμούσαν εδώ να είχαν περισσότερο χρόνο για να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Ε, try Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να, προσπα... και να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω από την τελευταία παρατήρηση. Η μελέτη αυτή έχει γραφτεί στο πνεύμα του εμπορίου, προσφέρει πολλές δυνατότητες. Δεν είναι μελέτη κατά του εμπορίου, είναι όμως μελέτη που εξετάζει πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη του εμπορίου και πώς μπορούν να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες ε, στην απασχόληση και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ε, δημόσια υποστήριξη για το εμπόριο. Αυτό είναι το πνεύμα ε, της μελέτης αυτής. Εγώ εργάστηκα 9 χρόνια για το ΠΟΕ και γι' αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να υιοθετήσω προστατευτικά μέτρα να αποδεχτώ προστατευτικά μέτρα. Να πάω σε μία από τις πρώτες ερωτήσεις. Οι πιο φτωχές χώρες ε, δεν έχουν πληγή. Ε, ναι, οι πλούσιες χώρες έχουν ε, επηρεαστεί περισσότερο διότι χτυπήθηκαν από δύο κρίσεις, την χρηματοοικονομική και την εμπορική. Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν πληγεί από την χρηματοοικονομική κρίση. Τι έγινε στις χώρες αυτές. Ε, τα στοιχεία τα βλέπετε όλα στην έκθεσή μας, αλλά για τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες σε χώρες όπως είναι η Λιβερία. Ε, το, μέχρι το 90% των θέσεων απασχόλησης ε, είναι στην άτυπη οικονομία. Έχουμε ε, κάποιες συνεντεύξεις ε, που έγιναν. Ξέρουμε ότι κάποιοι έχασαν το 80% του οικογενειακού εισοδήματος. Ξέρουμε ότι ο κόσμος ε, αγωνίζεται να επιβιώσει επειδή δεν έχει εισόδημα, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν είναι επιστημονικές. Γι' αυτό είναι δύσκολο να λύσουμε τέτοιου τύπου στοιχεία. Η παγκόσμια κοινότητα λοιπόν, ο ΔΟΕ, μπορεί να, να, βοηθήσει βρίσκοντας περισσότερες πληροφορίες και στηρίζονται στηρίζοντας ε, πρωτοβουλίε για να συλλεχθούν καλύτερα στοιχεία όχι μόνο όσον αφορά τον αριθμό, την ε, ποσότητα των ε, θέσεων αποσχόληση, αλλά και την ποιότητα, δηλαδή τι αμοιβέ. Θα πρέπει να εργαστούμε πιο ενεργά για την ε, ποιότητα και την ποσότητα των θέσεων απασχόλησης ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιες ε, νέε ρήτρε. Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να απαντηθεί από αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική. Μπορώ να σας πω όμως τι κάνει αυτή τη στιγμή η ΔΟΕ. Πρόσφατα γίναμε μέλος του κλάστερ των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και το παραγωγικό δυναμικό. Ε, έτσι λοιπόν ε, μαζί με, άλλες, ε, μαζί με άλλους φορείς ασχολούμαστε με προγράμματα που σχετίζονται με το εμπόριο. Προσπαθούμε να κάνουμε το εξή. Προσπαθούμε να κάνουμε τι χώρες ε, πιο ανταγωνιστικέ, ε, ε, παράλληλα όμως δίνοντα προσοχή στι συνθήκε της απασχόληση και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τι χώρες να αναβαθμίσουν την ποιότητα των εξαγωγών του. Έτσι μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ και να εξάγουν, αλλά θέλουμε παράλληλα να πληρώνουν σωστού μισθού και να παρέχουν καλέ θέσει απασχόληση. Το θέμα είναι λοιπόν πώς μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές ε, έχοντας καλές συνθήκες. Η παραγωγικότητα συχνά αυξάνεται όταν είναι καλύτερες συνθήκες εργασίες. Ε, βελτιώνεται η ποιότητα των ε, θέσεων απασχόλησης, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Θέλουμε επίση να βοηθήσουμε τι χώρε να διαφοροποιήσουν περισσότερο τι οικονομίε του και την παραγωγή του για να είναι λιγότερο ευάλωτε σε κλονισμού. Η δουλειά που κάνουμε λοιπόν ε, μπορεί να βοηθήσει τον ΔΟΕ να ε, βοηθήσει τις χώρες να είναι λιγότερο ευάλωτες ε, στους εξωτερικούς κλονισμούς. Άλλος τομέα στον οποίο εργάζεται η ΔΟΕ είναι η παροχή κοινωνικής προστασίας. Να βοηθήσουμε δηλαδή τις χώρες να οικοδομήσουν ε, την κοινωνική τους προστασία, να ε, βελτιώσουν το δυναμικό τους, ε, να βελτιώσουν συστήματα προστασίας σε διάφορες χώρες, διότι το ποια είναι η σωστή κοινωνική προστασία εξαρτάται από πολλά πράγματα και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η υποστήριξη λοιπόν αυτών των πρωτοβουλειών είναι κάτι που επικροτούμε ιδιαίτερα. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας δώσω πληροφορίες για ένα άλλο πρόγραμμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι κοινό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και έχει αντικείμενο ένα βιβλίο που ονομάζεται «Παγκοσμιοποίηση ε, κοινωνικά βιώσιμη». Ε, ασχολούμαστε με τη δημιουργία θέσεων αποσχόλησης και το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται από τους δύο φορείς που συμμετέχουν Στόχος μας είναι να δούμε πώς μπορεί η παγκοσμιοποίηση να ε, λειτουργεί προς όφελος όρων. Έχω πολύ λίγα ε, αντίτυπα του βιβλίου. Σύντομα θα είναι προσπόληση μέσω του διαδικτύου ή και σε βιβλιοπολία. Αυτή τη στιγμή τα βιβλία έχουν κολλήσει κάπου ανάμεσα στην Ινδία και την Γενέβη επειδή ε, χρησιμοποιήσαμε το τοπικό, ε, την τοπική αλυσίδα προμήθειας ε, για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί κόσμος θα έχει πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορούν να επανέλθουν σε εσά. Θα ήθελα να κλείσω την συνεδρίαση. Έχουμε ξεπεράσει λίγο το χρόνο μας. Η πρόεδρο, ζητεί συγγνώμη από του διερμηνείς. Ε, κυρία Γιάνσεν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Μορέιρα, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, 9 η ώρα, αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε και θα ξεκινήσουμε με την ε, ανάπτυξη του... Ε, ε, με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργία θέσεων εργασία στο πλαίσιο μια βιώσιμη οικονομία. Ευχαριστώ.